Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε Επίτροπε. Θα αρχίσουμε τώρα την συζήτηση και εξ ονόματος του Λαϊκού Κόμματος πρώτος λαμβάνει το λόγο ο κύριος Μπάλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλόρδε Χίλ. Δύο σύντομες ερωτήσεις που νομίζω ωστόσο έχουν γενική σημασία. Αφενός, τα πιστοτικά ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακρίνονται κατά μέγεθος, περιπλοκότητα κτλ. Ενίοι κανόνες και τεχνικές προδιαγραφές καθιστούν για μικρές και μεσές επιχειρήσεις συχνά δύσκολο να προωθούν τα επιχειρηματικά τους πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ασκεί την αναλογικότητα. Αυτή τη ρήτρα της αναλογικότητας πρέπει βέβαια να της εμφυσιθεί ζωή. Γι' αυτό θα ρωτήσω, ως μελλοντικός επίτροπος, πώς θα εξασφαλίσετε αυτή η αναλογικότητα να μην χρησιμοποιείται ως εξαίρεση, αλλά να γίνει ο κανόνας. Αυτή ήταν η, η πρώτη ερώτηση. Δεύτερο, μελέτη επιπτώσεων για την συσσόρευση των πολιτικών της ενιαίας αγοράς κανονισμών και οδηγιών. Ως μελλοντικός επίτροπος πώς θα προχωρήσετε σε μια τέτοια μελέτη. Κύριε υποψήφιε. Σας ευχαριστώ κύριε Μπάλτς. Νομίζω ότι θίξατε δύο πολύ σημαντικά θέματα. Πώς θα εξασφαλιστεί η ισορροπία σε ό,τι αφορά την νομοθεσία και πώς θα εξασφαλίσει κανείς επίσης ότι σε όλο το ευρώς θα έχουμε νομοθεσία αναλογική και ότι μπορούμε να παρακολουθούμε επίσης και τις επιπτώσεις που έχει στους διάφορου τομείς. Όσον αφορά την αναλογικότητα, η απάντησή μου μπορεί να είναι ότι σε αυτήν θα επανέλθουμε βέβαια, αλλά είναι η σημασία μιας ισορροπίας. Ασφαλώς χρειαζόμαστε νομοθετικές ρυθμίσεις που να λειτουργούν. Δεν θα πρέπει ωστόσο να θεωρήσουμε ότι κάθε επιχείρηση έχει το ίδιο μέγεθος και γι' αυτό ότι χρειάζεται μια προσέγγιση του είδους one size fits all. Σημειώνω λοιπόν το επιχείρημά σας για την αξία της αναλογικότητας. Σε ό,τι αφορά τώρα την προσπάθεια υπολογισμού των επιπτώσεων της νομοθεσίας συνολικά, νομίζω ότι αυτό πράγματι είναι πολύ σημαντικό και εφόσον επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου, θα το αναπτύξω. Σε διάφορες συζητήσεις που διεξήγαγα με μέλη της Οικονομικής Επιτροπής από διάφορες πολιτικές ομάδες, μου έθεσαν υπόψη τα μέλη αυτά ότι θα είναι χρήσιμο να έχουμε μια συνολικότερη προσέγγιση για το σωρευτικό αποτέλεσμα της νομοθεσίας σε διάφορους τομείς. Ενστικτοδός θεωρώ ότι πράγματι αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να το αντιμετωπίσει κανεί. και μία από τις προκλήσεις της νομοθεσίας και εγώ βέβαια θα χρειαστεί πρώτα να ενημερωθώ για αυτό τον περίπλοκο τεχνικά τομέα, είναι ότι υπάρχουν μεγάλα ποσά δραστηριοτήτων σε πολλούς τομείς και κλάδους και θα πρέπει να δω, να δω ποια είναι η επίπτωση του ενός τομέα στον άλλο. Αυτό θα χρειαστεί να κάνω βεβαίως εφόσον ευαιωθεί ο διορισμός μου. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ελίζα Φερέιρα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στα αγγλικά για να διευκολύνω το διάλογό μας. Σας ευχαριστώ που προσήλθατε ενώπιόν μας, κύριε υποψήφια επίτροπε. Στις γραπτές σας απαντήσεις λέτε ότι δεν μπορείτε να δεσμευτείτε μονομερός για πρόταση οποιασδήποτε πρωτοβουλίας. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή το όργανο στο οποίο επιθυμείτε να ενταχθείτε, δραστηριοποιείται στην δημιουργία της Τραπεζικής Ενώσεως σε επικοδομητική συνεργασία με την Ευρωβουλή, όπως τα έχετε δει κι εσείς. Αυτή η Τραπεζική Ένωση βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Έχουμε τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, έχουμε και τον ενιαίο μηχανισμό επίλυσης και το τελευταίο κομμάτι που μένει είναι ο τρίτος πυλώνας. Είναι η κοινή εγγύηση καταθέσεων που εφόσον δεν υπάρξει λείπει ένας σύνδεσμος. Ερώτηση λοιπόν, θα μας υποβάλλετε πρόταση για ενιαίο σύστημα εγγύησεως καταθέσεων που είναι το εναπομένον κομμάτι του puzzle. Θα το κάνετε πριν από το τέλος του 2015 και ποια θα είναι η δομή του ε, προγράμματος αυτού. Κύριε υποψήφιε, ευχαριστώ και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να θίξω το σημαντικό θέμα της Τραπεζικής Ενώσεως που αποτελεί κέριο τμήμα των καθηκόντων που ενδέχεται να αναλάβουν και όπως είπατε και πρώτη στην προτεραιότητα βεβαίω είναι να μπει το επόμενο κομμάτι του puzzle. Δηλαδή πρώτα να βεβαιωθούμε ότι διαθέτουμε τα κατάλληλα μέτρα για να, έχουμε, να λειτουργήσει το ενίο, το ταμείο για την διάλυση και αυτό θα το κάνω και στη βάση ρυθμίσεων backstop. Σε ό,τι αφορά το σύστημα ε, εγγύησης καταθέσεων, γνωρίζω ότι αυτό συζητείται εντονότατα τους τελευταίους μήνες και εδώ στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά είμαι σίγουρος και γενικότερα. Και νομίζω ότι η προσέγγιση που θα επιλέξω θα είναι ότι προτεραιότητα για μένα θα είναι να εφαρμόσω τη διαδικασία ως προβλέπεται τώρα η προσέγγιση δηλαδή που έχει επιλεχθεί και σε ό,τι αφορά τη γενικότερη συζήτηση, αν θα καταθέσω δηλαδή πρόταση πριν από το τέλος του έτους, δεν νομίζω ότι μπορώ να σας υποσχεθώ τώρα, αλλά όταν θα έχω προχωρήσει με την προσέγγιση που ήδη ισχύει, θα δω πόσο θα έχει προχωρήσει το σύστημα εγγυήσεω καταθέσεων. Νομίζω ότι αυτή είναι και η συνήθι προσέγγιση άλλωστε. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα συζητήσουμε ξανά στον χρόνο που έρχεται και αυτή θα είναι και η προσέγγιση μου. Σας ευχαριστώ. Swinburne, ECR. Ευχαριστώ, Μιλόρδε Χιλ αγγλικά θα μιλήσω μαζί σας, όχι ουαλικά, μην ανησυχείτε. Θα σας ερωτήσω ορισμένα πράγματα για τις αγορές, αλλά καλύτερα αργότερα αυτά. Δοθέντος ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες από τότε που κατέστη γνωστή η υποψηφιότητά σας, παρακολουθώ στους διαδρόμους τα τεκτενόμενα και κάτι το οποίο τίθεται ξανά και ξανά είναι σχετικά με το βιογραφικό σας και ιδίω ότι δύο γνωστές εταιρείες, γνωστές εδώ, Label Communications και Label Pottinger Communications, εμφανίζονται στο βιογραφικό σας. Και μάλιστα εσείς έχετε κάνει και μια εταιρεία που λέγεται Quiller Consultants. Θα είναι σημαντικό για μας να αναπτύξετε το θέμα αυτό ανοιχτά και να εξηγήσετε τον ρόλο σας μέσα στις εταιρείες αυτές και να εξηγήσετε κιόλας εάν διαθέτετε ακόμα κάποια συνεχιζόμενη σχέση με τις εταιρείες αυτές. Ο κύριος Χίλ, χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να θίξω το θέμα, ιδίω για την Quiller Consultants, που είναι η business την οποία ξεκίνησα εγώ το 1998, γιατί τις άλλες δουλειές αυτές είναι πριν από 25 περίπου χρόνια και ε, βέβαια η μνήμη μου δεν είναι η ίδια που ήταν τότε. Σε ό,τι αφορά τη δική μου δουλειά, χαίρομαι. Είμαι υπερήφανος που την ξεκίνησα από το μηδέν. Κατάφερα να προσλάβω και ανθρώπους πληρώσαμε φόρους, προσφέραμε απασχόληση και παρόλο που την ε, πούλησα προκταετίας και έφυγα εντελώ πριν από 4,5 χρόνια, συνεχίζει να υπάρχει η εταιρεία αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα το άτομό μου και οποιαδήποτε σχέση μπορεί να έχω με την εταιρεία αυτή, όταν μου ζητήθηκε να μπω στην Βρετανική κυβέρνηση ως Υπουργό Παιδείας, έτσι λειτουργούν στη χώρα μου τα πράγματα αυτά, έφυγα από την εταιρεία μέσα σε λίγες ώρες. Και αυτό υπήρξε και το τέλος οποιοδήποτε δεσμού είχαμε αυτήν. Είχα κάποιες μετοχές της εταιρείας αυτής που μου είχαν δώσει τότε που την πούλησα. Τότε τις είχα αποκαλύψει όταν ήμουν Βρετανός υπουργό, όταν διορίστηκα επειδή δεν ήθελα κανείς να σκέπτεται ότι υπάρχει κάποιο ίχνος συγκρούσεως συμφέροντος, έδωσα οδηγίες μέσα και σε λιγότερο από μια μέρα από τη στιγμή που διορίστηκα να φύγουν οι μετοχές αυτές, κάτι το οποίο έγινε μάλιστα ταχύτατα. Πολύθηκαν λοιπόν, έφυγαν και νομίζω ότι σύγκρουση συμφερόντων όντω είναι ένα κέριο θέμα που όλοι πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Νομίζω το κλειδί για την σύγκρουση συμφερόντων είναι πιο πολύ υπάρχει περίπτωση κάποιος να υποφεληθεί από κάποια απόφαση που θα λάβει ως επίτροπος, είτε επειδή έχει μετοχές, είτε επειδή βρίσκεται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάποιας εταιρεία. Και στις δύο αυτές τις περιπτώσεις η απάντηση είναι όχι, όχι και όχι. Άλτε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ το, ε, ευχαριστώ κύριε Χίλ. Θα μιλήσω αγγλικά όχι για να σα κριτικηθώ για τη χρήση σα του λόγου του Μολιέρου, της γλώσσα του Μολιέρου, αλλά για να εξυπηρετήσω. Λέτε στη δήλωσή σα ότι για την τραπεζική αρχή και τη λήψη αποφάσεων εκεί όπου απαιτείται η πλειοψηφία και από τον ε, κοινό εποπτικό μηχανισμό και τι αρχέ του και από τα 28 κράτη-μέλη, λέτε και παραθέτω ότι όλοι οι νόμοι φαίνεται να λειτουργούν σωστά χωρίς να εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού λήψης αποφάσεων. Μπορείτε να δεχτείτε την συνέχιση, την ευρύτερη εφαρμογή ενός συστήματος που κατά τη γνώμη μου δημιουργεί κενά ή κατακαιρματισμό στην ενιαία αγορά και δίνει κάποια δικαιώματα βέτο κυρία σε κάποια κάτι μέλη. Με συγχωρείτε πρώτα απ' όλα για όσα έκανα στη γλώσσα του Μολιέρου στις ε, προκαταρκτικές μου παρατηρήσεις. Λυπούμε πραγματικά και ζητώ συγγνώμη από τους Γάλλους ομιλητές. Τώρα, ε, για την ουσία της ερώτησής σας. Οι συγκεκριμένες διευθετήσεις που ισχύουν και που έγιναν δεκτές όταν ασχοληθήκαμε με την Τραπεζική Ένωση προέκυψαν από κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες εκείνο τον καιρό. Αυτές ισχύουν ακόμα εξ όσων γνωρίζω και από τις πληροφορίες που έλαβα και από ό,τι ξέρω λειτουργούν εύρυθμα. Η απάντησή μου στην ερώτησή σας θα είναι αρκετά σύντομη. Εάν το βλέπω αυτό ένα πρότυπο που θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Νομίζω ε, το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε για τις συγκεκριμένες συνθήκες, για τις ανάγκες της Τραπεζικής Ένωσης. Η σχέση για να μπορέσει να καλυφθεί η σχέση όσων συμμετέχουν και όσων δεν συμμετέχουν. Ευχαριστούμε για την ΚΟΕ. Μαρτ Κάρτη. Κύριε Ψήφια Επίτροπε, τον Ιούνιο του 2012 το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, αποφάσισε να σπάσει αυτή τη σύνδεση μεταξύ του εθνικού και του ιδιωτικού ε, χρέους και η Ιρλανδική κυβέρνηση είδε ότι ένα κομμάτι των χρημάτων αυτών αφαιρέθηκε από τον Ιρλανδικό λαό για να σώσει το τραπεζικό σύστημα. Αυτό ίσως ε, να είναι κατάλληλο σε κάποιους, να φαίνεται κατάλληλο σε κάποιους, αλλά καταλαβαίνετε ότι για τους Ιρλανδούς 40% της κρίσης των τραπεζών πληρώθηκε από τον ίδιο τον λαό και θα είστε μέλος του Σώματος των Επιτροπών παρά το γεγονός ότι δεν θα είναι αυτό ακριβώς τον τομέα των αρμοδιοτήτων σας. Ερωτώ λοιπόν, θα υποστηρίξετε επί της αρχής σε ό,τι αφορά την Ισλανδία και άλλες κυβερνήσεις για την ανδρομική επανακεφαλοποίηση προκειμένου να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και προφανώς καταλαβαίνω πόσο σημαντικό και ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα για το λαό της Ιρλανδίας ε, στι δυσκολίες ε, που αντιμετώπισαν εκείνη την εποχή. Ξέρω επίσης ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο συζητήθηκε ε, εκτεταμένα σε όλο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής του, μου είπαν ότι από νομικής απόψή είναι δυνατόν να γίνει αυτό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού σταθερότητα για αναδρομική ε, επανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Και αυτό ισχύει. Πολύ φοβάμαι ότι εδώ δεν μπορώ να σας δώσω την ενθάρρυνση την οποία θα θέλατε. Οποιαδήποτε απόφαση όμως λοιπόν για το θέμα αυτό θα πρέπει να ληφθεί μετά από εξέταση κατά περίπτωση και προφανώς θα έπρεπε τα κράτη του Σευροζώνης να αποφασίσουν μια, να πάρουν μια τέτοια απόφαση με ομόφωνη βάση. Αλλά όπως σας είπα ο κύριος Μασκοβίτσι θα είναι ο καθήλυν αρμόδιος αν αυτό προταθεί σε κάποια φάση προφανώς θα είμαι τμήμα της ομάδας που θα εξετάσει το αίτημα αυτό και δεδομένης της κατάστασης και δεδομένης ε, της σύνθεσης. Είμαι σίγουρος ότι θα λεφτεί μια τέτοια απόφαση ενδεχομένω. Ευχαριστώ πολύ. Για τους πράσινους, ο Σβεν Γκίγκολτ. Λόρτε Χίλ, καλώς ορίσατε. από την διαπραγμάτευση της συνθηκών του έχει τη σχέση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει ψυχρανθεί από πολλές απόψεις. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ευρωπαϊκή σας δέσμευση. Εσείς ο ίδιος, τι έχετε πράξει, τι έχετε κάνει ως δημόσιο άτομο, ως προσωπικότητα εκείνη την εποχή και σε αυτές τις εποχές προκειμένου να ενισχύσετε τη σχέση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος. Επίσης, μία άλλη ερώτηση. 200.000 λομπιίστες και εργάζονται εδώ στις Βρυξέλλες. Το City of London Corporation καλωσορίζει την υποψηφιότητά σας και εσείς έχετε ιδρύσει στο παρελθόν μία τέτοια εταιρεία λομπιίστων. Αναρωτιέμαι, μήπως ε, βάζουμε τον ελέφαντα μέσα στο κατάστημα με τις πορσελάνες. Αναφερθήκατε ιδιαίτερο σε θέματα διαφάνειας. Για ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχετε εργαστεί εσείς ή οι εταιρείε σας, θα ήθελα να ξέρω. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη δέσμευσή μου για το να διαδραματίσει η Βρετανία ενεργό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο ήθελα να πάρω τη δουλειά αυτή και για τον οποίο ήρθα εδώ πριν από 25 χρόνια. το 1 τέταρτο του αιώνα δηλαδή, κατά τη διαπραγμάτευση της συνθήκη του Μάστρεχτ, ήμουν στην ε, Πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας και πριν ε, δούλεψα για τον Γκένεθ Κλάρκ. Άρα η εμπλοκή μου και η δέσμευσή μου σε ευρωπαϊκά θέματα και η κατανόηση της σημασίας και της πολιτικής ευαισθησίας του στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάτι το οποίο έχω ζήσει στο πετσί μου 25 χρόνια. Είναι σαφείς και ξεκάθαρες οι απόψεις μου. Ελπίζω ότι τις ε, παρουσίασα σωστά που είναι ότι είναι υπέρ του συμφέροντος της ε, Βρετανίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά για την πρώτη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη ερώτηση τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις μου. Ξεκίνησα Αναφερόμενο σε τέτοια θέματα στην εισαγωγή μου να τονίσω και πάλι ότι έφυγα πριν από 4,5 χρόνια από την επιχείρηση τρεις φορές δηλαδή το, η περίοδος που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορεί να θεωρηθεί κάποιος αμερόληπτος και να αναλάβει σχετικά καθήκοντα. Είναι πάρα πολύ σωστό που υπάρχει αυτή η περίοδος που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί καταλαβαίνω και το άγχος του κόσμου, την ανησυχία των πολιτών ότι μπορεί να έρχεται ο κόσμος να αναλαμβάνει καθήκοντα α, πολιτικά προς το δικό του συμφέρον. Δεν είναι αυτός ο λόγος που ήρθα εδώ σήμερα για να κάνω τη δουλειά αυτή. Δεν έχω καμία ιδέα για το τι θα μου φέρει το μέλλον και δεν είμαι εδώ ως εκπρόσωπος του City του Λονδίνου. Είμαι εδώ ελπίζοντας να μπορέσω να εκπροσωπήσω τους Ευρωπαίους και να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις σε ό,τι αφορά τη σωστή νομοθεσία και την σταθερότητα, ελπίζω και την ανάπτυξη προς όφελος όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ακολουθήσω την επιχειρηματολογία, τη λογική της νομοθεσίας για να το εφαρμόσω αυτό σε διασυνοριακό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Good morning, Lord Hill. So pleased to hear Καλημέρα σας, Λόρδε Χιλ. Χαίρομαι που ακούω μια φωνή Βρετανού μια τόσο από μια τόσο υψηλή θέση. Κάτι σπάνιο σε αυτό το κτίριο. Στο διορισμό σας στην ε, Βουλή, ως μέλος της Βουλής των ε, Λόρδων. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Ε, ως στο διορισμό σας στην Βουλή των Λόρδων ορκιστήκατε ενώπιον της ε, Βασιλισσάς ότι θα είσαστε πιστός μόνο στην υψηλότητά της. Εάν εγκριθείτε έναν παρόμοιο όρκο θα δώσετε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είστε τελείω ανεξάρτητο στην ε, ε, διεξαγωγή των καθηκόντων σα και προ συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί να λαμβάνετε οδηγίε ή ε, να παρενοχλήσετε από οποιαδήποτε κυβέρνηση, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, φορέα ή οντότητα, νομική οντότητα. Σίγουρα ε, μεταξύ σα οι δύο όρκοι. Όπω λέγεται και στην ε, βίβλο του, ε, βασιλιά, του King James. Ε, κανένας άντρας δεν μπορεί να, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να, είναι υπηρέτης δύο αφεντάδων. Ποιος είναι τώρα ο αφέντης σας, η Βασίλισσα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην προηγούμενη δουλειά μου, ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια ως ε, σύμβουλος και ως υπεύθυνο για το Λάγκαστέν ήταν να συναντήσω την ίδια την ε, Βασίλισσα. Αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Ουδέποτε πίστεψα, ούτε για μια στιγμή, ότι η ψηλότητά της θα θεωρήσει ότι ο όρκος που ορκίστηκα μπροστά της θα αντιφάσκει με τον όρκο που θα μπορέσω να ορκιστώ εδώ, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου ως Επιτρόπου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία αντίφαση. Ευχαριστούμε από τους ε, μη εγγεγραμμένους Γκέρολφ Άνεμανς. Με συγχωρείτε, αλλά παραβαίνει ένα πολιτικό ερώτημα, κύριε Χίλ. Γιατί δεν αναλάβατε την αλία ή κάτι τέτοιο ως επίτροπος. Και το σίδι του Λονδίνου βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί σας διάλεξε εσάς ο Γιούνκερ για τη χρονοτοποστατική σταθερότητα και την Ένωση των Κεφαλοχικών Αγορών. Γιατί επέλεξε γι' αυτό τον Βρετανό υποψήφιο. Η απάντησή σας ότι το, κάποια στοιχεία θα τα καλύπτει ο κ. Ντομπρόφσκης δεν επιλύει την αντίφαση. Το θέμα είναι η οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης και αυτό το αδιέξοδο το οποίο έχει φέρει το ευρώ τις οικονομίες των μελών του. Οι ευρωσκεπτικιστές και το συντηρητικό σας κόμμα και το Ηνωμένο Βασίλειο γενικώ έχουν δίκιο όταν δηλώνουν ότι η Ένωση δεν πρέπει να γίνεται σε λάθος βάσης. Για τη δική σας λοιπόν την περίπτωση υπάρχει σαφώς ε, μια ε, αντίφαση μεταξύ της Ένωσης των Χρηματοπιστωτικών Αγορών και το να θέλετε να παραμένετε εκτός οποιοδήποτε κοινού νομίσματος ή Χρηματοπιστωτικής Ένωσης ή Δημοσιονομικής Ένωσης. Για το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, γιατί προτάθηκα για το χαρτοφυλάκιο αυτό, αυτή είναι μια απόφαση που έλαβε ο κύριος Γιούνκερ. Ε, ήταν, ήμουν, τιμή μου να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Είναι πολύ σοβαρές οι ευθύνες που θα αναλάβω και θα φροντίσω να τις φέρω εις πέρας κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν δέχτηκα αρχικά τον διορισμό από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, δεν ήξερα ποιο χαρτοφυλάκιο θα αναλάβω προφανώ. Θα μπορούσα να είχα καταλήξει στην Αλία, αλλά ανέλαβα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τον κανονισμό για την Ένωση των Κεφαλογικών Αγορών. Αυτό μου ζητήθηκε να αναλάβω. Νομίζω όμως ότι εδώ έχουμε μία εκδοχή, τέλος πάντων μια διαφορετική εκδοχή της προηγούμενης ερώτησης για τις εντάσεις και πώς μπορεί κανείς να τις καταπραίνει νομίζω ότι θα είναι προς όφελος και των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ευρώ να είναι επιτυχημένο και να μπορέσει να ανθίσει, να ευδοκιμήσει. Νομίζω ότι είναι προς όφελος και των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πετύχει η Τραπεζική Ένωση. Και βεβαίως να είναι ανοιχτή δεχτεί η Τραπεζική Ένωση σε οποιοδήποτε από τα 28 κάτι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και αν δεν είναι μέλη τη Ευρωζώνη, να μπορούν να συμμετάσχουν στην Τραπεζική Ένωση. Βεβαίω έχω μιλήσει με πολύ κόσμο τι τελευταίε εβδομάδε για τα θέματα αυτά και όντω υπάρχουν τριγμοί και εντάσει σε πολλά θέματα όμω, αυτό που συλλογικά έχουμε να λάβει ω ευθύνη, αν μου επιτρέπετε, είναι να προσπαθήσουμε να καταπραίνουμε, να διασκεδάσουμε τι αμφιβολίε και να καταπραίνουμε τι εντάσει. Και για παράδειγμα στην Τραπεζική Ένωση να ε, έχουμε τον ενιαίο, τους ενιαίους κανόνες για όσους είναι μέλη της Ευρωζώνης όπως και για όσους δεν είναι. Ακολουθεί ο κύριος Χεκμαρκ. Σας ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επιτροπέ. Το Ενωμένο Βασίλειο είναι σημαντικό τμήμα μιας ισχυρής ε, Ενωμένης Ευρώπης παγκόσμια και ελπίζω να παίξετε και εσείς ένα σημαντικό ρόλο. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα, πώς βλέπετε τον συντονισμό και την ε, διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ ημών του κ. Μοσκοβισή και του κ. Κατάινεν. Πώς θα διακρίνετε ποιος είναι αρμόδιος για ποια πράγματα και πώς θα διασφαλίσετε αποτελεσματικότητα καθώς και αποτελέσματα συνέργειας στην συνεργασία σας. Δεύτερο, όλοι μιλούν για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών και λίγοι μπορούν να εξηγήσουν τι ακριβώς είναι. Πώς θα τα καταφέρετε. Δηλαδή, οι ευρωπαϊκές αγορές είναι κατακαιρματισμένες. Και γι' αυτό και δεν αποδίδουν στο μέγιστο του συνόλου των ικανοτήτων τους και όχι μόνο οι χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά και ολόκληρη η οικονομία. Πώς θα καταφέρετε λοιπόν να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πρώτα για το σημαντικό θέμα του συντονισμού που θίξατε. Η άποψή μου είναι πρώτα ότι η ιδέα να υπάρξουν ομάδες επιτρόπων που θα συνεργάζονται, που θα συντονίζονται και που θα τους ενθαρρύνει ένας αντιπρόεδρος της Επιτροπής, νομίζω ότι είναι καλή η ιδέα αυτή. Είναι καλό που γίνεται η προσπάθεια να γίνει αυτή η ομαδική προσπάθεια από έναν αριθμό επιτρόπων, εφόσον υπάρχουν αλληλοσυνδεόμενα θέματα, νομισματική ένωση και σχετική ε, νομοθεσία, ανάπτυξη και απασχόληση που μπαίνει και σε άλλα χωράφια και νομίζω ότι έχει πολύ νόημα να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κοινή προσπάθεια. Είμαι λοιπόν υπέρ της ιδέας αυτής. Τώρα, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ξέρω ότι ο jean Κλοντ Γιούνκερ σε επιστολή προς τον πρόεδρό σας Μάρτιν Σούλτς έχει σκιαγραφίσει τις διάφορες αρμοδιότητες που θα έχουν οι αντιπρόεδροι. Η δική μου ε, απάντηση βασισμένη στην κοινή λογική είναι ότι πολλά θα εξαρτηθούν και από την προσωπική σχέση που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στους επιτρόπους. Εγώ πάντως θα μπω στην υπόθεση αυτή με αποφασιστικότητα να συνεργαστώ με τους κυρίους Μοσκοβισή, Κατάινεν, Ντομπρόφσκης. Είμαι λοιπόν πολύ υπέρ αυτής της προσεγγίσεως. Υπάρχει ένα κέριο θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι το ζήτημα της λογοδοσίας, accountability. Πρέπει να είναι σαφές ποιος θα λογοδοτεί ενώ ποιον σας. Ποιος θα έρχεται να σας εξηγεί. Πάντω, επαναλαμβάνω ότι είναι κέριο γι αυτό, αυτό για μένα. Βλέπω ότι θα με διακόψει ο πρόεδρο για τι κεφαλαιοαγορέ και την Ένωση των ε, Κεφαλαιογορών. Ε, ε, ελπίζω ότι κάποιο άλλο θα ρωτήσει και θα μπορέσω να απαντήσω ταυτόχρονα και σε εσά. Ευχαριστώ. Ιάκωβος Φον Βάιτσέκερ. Ευχαριστώ. Δεν θα σα ρωτήσω γιατί σίγουρα αφού υπήρξατε Σύμβουλο και του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα στο παρελθόν. Δεν θα σα ρωτήσω ποια συμβουλή θα δίνατε στον κύριο Γιούνκερ για την κατανομή των χαρτοφυλακίων. Θα σα ρωτήσω μάλλον για την Τραπεζική Ένωση και τις σχέσεις με τις χώρες εκτός Τραπεζικής Ένωσης, διότι η κρίση κατέδειξε ότι η νομοθετική συνεργασία είναι μια υπόθεση όταν τα πράγματα πάνε καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οδηγηθεί σε όλο και αυστηρότερες εξοδαφικές ρυθμίσεις για τράπεζες που υπάρχουν και σε άλλες δικαιοδοσίες. Θα υποστηρίξετε το ίδιο αυστηρές ρυθμίσεις για τις εθνικές επιχειρήσεις εκτός των, ε, του χώρου εφαρμογής της Τραπεζικής Ένωσης. Ή αυτό που είπατε θα γυρίσετε τηλεσκόπιο ανάποδα για να έχετε τη μακρό ε, άποψη θα οδηγήσει την πραγματικότητα σε μια διάχυση της προσπάθειας. Για το πρώτο σας θέμα. Ο Ζαν και ξέρει πολύ καλά τι θέλει και δεν έχω καμιά συμβουλή να του δώσω. Τώρα για την ουσιαστική σας ερώτηση, για την Τραπεζική Ένωση, για τους in και για τους out και όλα τα σχετικά. Αξίζει τον κόπο να θυμίσω και πάλι Γνωρίζω βέβαια ότι πολλοί είναι ευαίσθητοι για τις ενδεχόμενες εντάσεις και για το γεγονός ενδεχομένως ότι εγώ είμαι υπήκος μιας χώρας που δεν συμμετέχει στην Τραπεζική Ένωση και έχουν λοιπόν αμφιβολίες για το αν θα είμαι ικανός να παίξω τον ρόλο, που εγώ πιστεύω ότι θα μπορέσω να τον παίξω τον ρόλο αυτό, διότι θα λειτουργήσω προς το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Υπάρχει λοιπόν το Single Rule Book, ενιαίοι κανόνες που δεσμεύουν και τι 28 χώρε μέλη και καλό είναι να τις θυμόμαστε αυτό. Και σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτησή σας για την εξοεδαφικότητα, νομίζω ότι όντω συμβαίνει αυτό. Ορισμένες φορές οι ΗΠΑ προσπαθούν να ρυθμίζουν τις τραπεζέ τους και παγκοσμίω, ακόμα και όταν είναι στην Ευρώπη. Το ερώτημά μου είναι εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις ΗΠΑ να τους πείσουμε να δεχθούν ως ισότιμους και τους κανόνες των άλλων. Αυτή είναι όμως και η ευρύτερη κρατούσα γνώμη και στο G20 και εγώ θα συνεργαστώ πάντως και με άλλους και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιτύχουμε αυτή, την εφαρμογή αυτή της αρχής και να μετριάσουμε έτσι τα προβλήματα που προβλέπετε εσείς. Μάλιστα ο αντιπρόεδρος μας Μάρκος Φέρμπερ. Ευχαριστώ, εγώ δεν θα μιλήσω ούτε τη γλώσσα του Σέξπιρου, του Μολιέρου, αλλά του Γκέτε, του Ιωάννου Βόλφκανγκ Φον Γκέτε, που αυτός μας έλειπε. Άμα θέλετε να σας τα λέω και στη διάλεκτο του Χέσεν όμως, κανένα πρόβλημα. Πρώτον λοιπόν, διαφάνεια. Είχατε δηλώσει ότι θα κοινοποιείτε όλες τις επαφές που έχετε και εκτός του Κοινοβουλίου. Τι έχετε να πείτε τώρα γενικά σχετικά με το νομοθετικό ίχνος. Θα μας τα πείτε όλα και Oxfam και City of London όλες τις σχέσεις ή επαφές που έχετε. Τώρα, ένωση των κεφαλαίων Αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται στην Ευρωζώνη, είναι μια παραπέρα εξέλιξη από την άλλη μεριά της ενιαίας αγοράς. Εγώ βλέπω δύο μεγάλα προβλήματα. Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Εκεί η ε, Ένωση των Κεφαλαιογόρων τι ρόλο μπορεί να παίξει σε αυτά τα δύο. Um, thank you for those, uh, three... Ευχαριστώ για αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Ως προς την ε, διαφάνεια, η προσέγγιση μου θα ήταν η εξής. Καταρχάς, να δω πολύ προσεκτικά την προσέγγιση του προκατόχου μου, ο οποίο φρόντιζε όλοι να γνωρίζουν τι συναντήσει είχε και αυτό θα το τηρήσω πιστά. Επίση, υπάρχουν προτάσει ευνοϊκές, προς τις οποίες είναι ευνοϊκές και ο κύριος Γιούγκερ να υπάρχει και ένα υποχρεωτικό μητρό για τα λόμπι που συναντούμε. Άλλωστε, οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον να συμμετέχει στην ε, χάραξη πολιτικής, οι ενώσεις καταναλωτών, οι πολίτες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Και με παρακολούθηση των χρηματοδοτικών εξελίξεων, οι πολίτες να ε, έχουν τι απαραίτητε πληροφορίε για αυτά τα τόσο τεχνικά ζητήματα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό και το παρακολουθούμε με προσοχή. Ω προ την Ένωση των Κεφαλαιγρών. Είμαι πολύ σαφή ω προ αυτό και ήταν το ίδιο και ο κύριο Γιούνκερ στην ανάθεση καθηκόντων και την επιστολή του προ εμένα. Αφορά και του 28 αυτό. Το εγχείρημα τη ενιαία αγορά ούτω ή άλλω αφορούσε του 28. Και δουλειά μου είναι να φροντίσω να αφορά και τους 28, ώστε να θέλουν να συμμετέχουν και τα 28 κρατη μέλη. Θα θεωρήσω ότι απέτυχα, εάν δεν είναι ένα κοινό εγχείρημα και για τα 28 κράτη-μέλη. Και πώς θα ενθαρρύνουμε τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ξέρω ότι υπάρχει μια σχετική πρόταση για την ενθάρρυνση των ε, σχετικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ε, Ένωση Κεφαλαίου Αγορών και για να προχωρήσει και θα φροντίσω να δοθεί προτεραιότητα σε, αυτό αυτή την πρόταση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Το σημειώνουμε αυτό που είπατε για το υποχρεωτικό μητρό διαφάνειας και τώρα λόγο στην κυρία Μπερές. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, στο κοινοβούλιο αυτό και επειδή χρειαζόταν μόγλευση και αντιμετώπιση της ε, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, επειδή θεωρήσαμε ότι χρειαζόταν ρύθμιση των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών και υπό την πίεση του συμπατριώτη σας, του κ. Μακάρθη, που επιχειρετίζω την ε, παρουσία στην αίθουσα αυτή, φροντίσαμε να δώσουμε κάποιες εγγύησεις προς τους τραπεζίτες το ίδιο όμω ήμασταν πολύ αποφασιστικοί για την πρόληψη τη χρήση του δημοσιονομικού χρηματοδοτικού συστήματο για τη λεύκανση προσόδων για την ε, χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Για λόγου σύγκρουση συμφερόντων, η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τα δύο αυτά κείμενα, δηλαδή η υπηρεσία Corporate Governance, δεν θα ανήκουν στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Το γεγονός ότι δεν θα μπορείτε να ασκήσετε αυτές τις αρμοδιότητες τελικά δεν σας καθιστά ανίκανο να μπορείτε να αναλάβετε τα θέματα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την Ένωση των Κεφαλαίων Αγορών. Um, uh, Πρώτον, για τη συγκεκριμένη ερώτηση, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το, αυτή είναι η εξήγηση. Η απόφαση που έλαβε ο κύριος Γιούνκερ ήταν τα θέματα αυτά να συστεγαστούν υπό την έννοια της ε, corporate governance. Τι καταλαβαίνω αυτή την ευαισθησία. Ως προς την ουσία όμως του θέματος, τα θέματα αυτά θα συζητηθούν στο σώμα των επιτρόπων, σε αυτό το επίπεδο και εκεί ελπίζω να διαδραματίσουν εργότατο ρόλο και φυσικά θα συνεχίσω να παρακολουθώ το θέμα. Πολύ σωστά πάντως είπατε ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σαφές ε, το τι θα συμβεί. Θα πρέπει να προχωρήσει η νομοθεσία και όπως κάθε επίτροπος θα πρέπει η νομοθεσία αυτή να εγκριθεί και να υλοποιείται. Η άποψή μου όμως για την ουσία του θέματος είναι ότι τα κίνητρα θα πρέπει να αντιστοιχούν στις επιδόσεις. Ένα από τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν είναι ότι αυτή η αντιστοιχία δεν ίσχυε πλέον κάποιοι δεν ε, λειτουργούσαν προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον των οργανισμών ή των ιδρυμάτων ε, για τα οποία δούλευαν, αλλά δούλευαν ε, προς όφελος των μετόχων. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο προκυπτούν προβλήματα. Για να λυθεί λοιπόν αυτό το πρόβλημα και οι σχετικές προτάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για το κλόμπακ ή για την ανάμιξη μετρητών με τίτλους, όλα αυτά για να φροντίσουμε να μην γίνονται σφαλμένες κινήσεις από όσους τα διαχειρίζονται είναι σημαντικό. Το τι θα γίνει όμως στη συνέχεια είναι κάτι που ακόμη και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξέρω ότι ο προκάτοχός μου παρακολούθησε το τι γινόταν με τις ε, αρχές των τραπεζών, τις ευρωπαϊκές αρχές τραπεζών και ζήτησε να συνεχίσουν την πορεία τους. Όμως όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα δημορφωθεί και η σχέση μας με την Eurover. Για την Επιτροπή ΙΜΚΟ τώρα, Ότμαν Κάρας. Καλώς ορίσατε, Λόρδε Χίλ. Θα ήθελα καταρχάς ε, να αναφερθώ στην επίστολη του κύριου Γιούγκρο, που αναφέρεται ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε την κοινωνική διάσταση και θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε ε, κίνητρα για τους μάνατζερ στις σχετικές υπηρεσίες, στις σχετικές βιομηχανίες. Πώς μπορείτε λοιπόν, πώς θέλετε να ανακτήσετε την κοινωνική δικαιοσύνη και πώς θέλετε να αποτρέψετε λανθασμένα μοντέλα. Δεύτερη ερώτηση. Η ενσωμάτωση, η ενοποίηση της ενιαίας αγοράς ε, σημαίνει ενοποίηση και της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Πού λοιπόν θα πρέπει να διαμορφωθεί η πιο ισχυρή και η πιο έντονη ε, ενοποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς για την έννοια της, εννοής, της ενιαίας αγοράς και ποια είναι, πιστεύετε, η σχετική απαραίτητη χρηματοδότηση και ποια σχέδια προτίθεστε να κάνετε για να χρηματοδοτήσετε εναλλακτικέ ε, μεθόδους τέτοιες. Για να ξεκινήσω από το τελευταίο σημείο. Πώς ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις στις αγορές. Νομίζω ότι με διάφορους τρόπους μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Το σημείο κίνησης μου για τις κεφαλαγορές και τις ενώσεις κεφαλαγορών θα ήταν να ξεκινήσω με μια προσεκτική και εις ανάλυση των ε, προσκομμάτων, των εμποδίων που υπάρχουν σήμερα σε ό,τι αφορά τις ε, σωστές και αποτελεσματικές ροές ε, κεφαλαίου σε όλη την Ευρώπη και μετά την ανάλυση αυτή να δούμε ποιες θα ήταν οι λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω δηλαδή, γιατί ξέρουμε ήδη ότι σε κάποια κράτη-μέλη θα υπάρχουν ε, διάφοροι που θα πούν ότι δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ σε άλλα κρατημέλη αυτό είναι έντονο πρόβλημα. Η συνολική, το συνολικό ζήτημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πολύ απλό ζήτημα του πώς θα υπάρξει καλύτερη αντιστοίχηση ενδεχόμενων επενδύσεων που έχουν παγώσει στην τρέχουσα φάση με τις επιχειρήσεις που χρειάζονται τις επενδύσεις αυτές για να αναπτυχθούν. Το πώς θα το πετύχουμε αυτό, όπως είπα και πριν από το Ταμείο Επένδυσης, ε, Μακροπρόθεσμος Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί ένα ε, ενδιαφέρον μοντέλο, που τα κονδύλια θα χορηγηθούν σε ε, έργα υποδομών, μικρομέσες επιχειρήσεις, επιστημονικούς κλάδους. Ενδιαφέρον λοιπόν είναι αυτό σαν μέθοδος Χρειάζεται και μία προσέγγιση που θα αυξήσει την ενημέρωση, γιατί ένα πρόβλημα με την κατακαιρματισμένη αγορά είναι ότι οι ενδεχόμενοι επενδυτέ δεν γνωρίζουν επαρκώ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει τι οποίε θα μπορούσαν να επενδύσουν. Άρα η πληροφόρηση είναι ένα βασικό ζήτημα. Τώρα, για αυτά που είπατε για τα κίνητρα για την κοινωνική διάσταση. Νομίζω ότι σε όλες μου τις δράσεις θα θέλαμε να σκεφτούμε ποια θα μπορούσαν να είναι τα ωφέλη για τους πολίτες της Ευρώπης και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν λανθασμένα κίνητρα που θα παροτρύνουν λανθασμένες συμπεριφορές. Ευχαριστώ πολύ. Φώτιγκαρ από το ECR, από τους συντηρητικούς και Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε υποψήφιε, ε, Επίτροπε, παρά το γεγονός ότι εν μέρει απαντήσατε στην ερώτησή μου ήδη, θα ήθελα να επαναλάβω κάτι από αυτά που είπατε εισαγωγικά. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ ευθέως. Πώς θα συμφιλιώσετε τα συμφέροντα των μελών της Ευρωζώνης και των χωρών που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Πώς θα εκπροσωπήσετε και τις δύο ομάδες επάξια. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο η πρόκληση που αντιμετωπίζω είναι η ίδια, αλλά αν θέλετε αντίστροφη σε σχέση με την πρόκληση που αντιμετώπισε ο κύριος ε, Μπαρνιέ. Οποιοςδήποτε βρίσκεται σε τέτοια θέση και εκτελεί τέτοια καθήκοντα, επειδή βρισκόμαστε στην παρούσα φάση εξέλιξης της Ένωσης, είναι είτε μέλος της ε, Ευρωζώνης είτε όχι. Ο Μισελ Μπαρνιέ είχε διοριστεί και τότε κάποιες ε, από τις χώρες που ήταν εκτός της Ευρωζώνης και ίσως και η δική μου χώρα ε, υποπτεύτηκαν και τον κατηγόρησαν ίσως ε, παράλογα ότι δεν θα ήταν σε θέση να συμφιλειώσει τα δύο καθήκοντα, τα δύο, τις δύο ιδιότητες αυτές. Και νομίζω ότι αποδείχθηκαν ε, λάθος, αποδείχθηκε ότι δεν είχαν δίκιο. Το ίδιο καθήκον έχω και εγώ, αλλά αντίστροφα θέλετε. Όπως λοιπόν ε, ο Μισελ Μπαρνιέ προσέγγισε τα καθήκοντά του από ευρωπαϊκής πλευράς, το ίδιο σκοπεύω να κάνω και εγώ. Πρακτικός πως τώρα για να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη, αυτό μπορεί να το πετύχουμε μέσω της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών, που θα πρέπει να αποτελεί μια ένωση των 28. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος να καταδείξουμε ότι είμαστε σε θέση να οικοδομήσουμε μια ενιαία αγορά προς το συμφέρον όλης της Ευρώπης, όπου και τα 28 κρατημέλη μπορούν να συμμετέχουν με ενθουσιασμό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό λοιπόν στις μελλοντικές μας εργασίες να έχουμε πάντα αυτό υπόψη και εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να φροντίσω ότι θα συμφιλειωθούν τα δύο αυτά συμφέροντα και θα συνενωθούν στην πολιτική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Νίον Χόιζεν από τους Φιλελεύθερους, η κυρία Νίον Χόιζεν από την ε, Φιλελεύθερους. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών. Αναφέρατε κάποια πράγματα για αυτήν, αλλά είναι λίγο νεφελώδες το τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε, σε ποιους κανονισμούς θα εστιαστείτε, τι θα πρέπει να αλλάξει. Αναφερθήκατε στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Συγκεκριμένα όμως, ποια είναι τα σχέδιά σας και πότε θα τα πετύχουμε. Σκοπεύετε να εισαγάγετε νέους κανονισμούς. Θα ήθελα περισσότερη, περισσότερες για τα θέματα αυτά. Γιατί στην παρούσα φάση είναι ένα ωραίο σλόγγαν. Α ενώσουμε τι κεφαλαγορέ. Αλλά τι ακριβώ σχεδιάζετε να κάνετε πέρα από τι καλέ προθέσει που αναμφισβήτητα έχετε και ακούσαμε. Απάντηση. Αυτό που λέω είναι το εξή. Το πρώτο βήμα λοιπόν, το οποίο ίσω να ακούγεται πολύ ε, κοινότυπο, αλλά είμαι πολύ πραγματιστή και ρεαλιστή, είναι ακριβώ να εντοπίσουμε ποια είναι τα εμπόδια, ποια είναι τα προσκόμματα για την ελεύθερη ροή των κεφαλαίων. Δεν θέλω να ξεκινήσω με, με μεγαλειώδη σχέδια και οράματα. Λίγο πριν από δύο εβδομάδες, ε, πριν από δύο εβδομάδες και ούτε καν ε, διορίστηκα. Νομίζω ότι θα ήταν παράλογο μετά από δύο εβδομάδες να έλθω και να σας πω ότι κοιτάξτε αυτά θα κάνουμε τα επόμενα πέντε χρόνια με λεπτομέρειες. Είναι σαφές λοιπόν στο μυαλό μου ότι θέλω βαθμιδών και σταδιακά να προχωρήσω. Όπως είπατε, υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου ήδη βλέπουμε ότι ενδεχομένως να χρειάζεται ε, κανονιστική ρύθμιση και νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανόν να χρειαστούν κανόνες για να αρθούν εμπόδια. Για το πώς, για παράδειγμα, μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις σε καλύτερη ποιότητα σε τιτλοποίηση αυτό ασφαλώς ε, πρέπει να το κάνουμε και ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο που να ξεκλειδώσουμε τις επενδύσεις χωρίς να διατρέξουμε τους κινδύνους που κανείς ε, δεν θέλει φαντάζομαι να διατρέξουμε. Άρα θα σας καλούσα κατεπηγόντως να δείξετε λίγη υπομονή γιατί νομίζω ότι θα ήταν ε, λάθος να βιαστούμε. Αλλά αυτό που είναι εντελώς ξεκάθαρο στο κεφάλι μου σε ό,τι αφορά την πρακτική εφαρμογή της Ένωσης Κεφαλαίου και του πώς θα άρουμε τα σχετικά εμπόδια είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα εντελεχώς να συζητήσω, να μελετήσω, να γίνουν διαβουλεύσεις και να χρησιμοποιήσω τις ιδέες όλων των εμπλεκομένων φορέων και της ΕΚΟΝ για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λούντιβιξον S&D, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, υποψήφια Επίτροπε. Δεν είναι ευκολότερη ίσω γλώσσα τα Σουηδικά. Πρόσφατα την Άνοιξη εγκρίθηκε νομοθεσία για την πρόσβαση σε έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Οι Ευρωπαίοι πολίτε ε, λέγεται ότι πλέον βάσει τη νομοθεσία μπορούν να αποτελούν τέτοιο λογαριασμό και κανεί δεν μπορεί να απορριφθεί από τι τράπεζε. Η Βρετανική κυβέρνηση όμω διαμαρτυρήθηκε. Δεν ήθελε να έχει τι ίδιε υποχρεώσει βάσει αυτή τη νομοθεσία και να δώσει τέτοια πλήρη δικαιώματα σε όλου του καταναλωτέ. Τώρα το νομοθέτημα αυτό έχει εγκριθεί και θα υλοποιηθεί στα κράτη-μέλη. Η ερώτηση μου λοιπόν προ εσά είναι εάν κάποια από τι κυβερνήσει των κρατών μελών προσπαθήσει να μην υλοποιήσει πλήρως ε, αυτό το νομοθέτημα. Τι θα κάνετε, θα το αφήσετε να συμβεί κάτι τέτοιο ή θα δείξετε πυγμή και θα φροντίσετε όλες οι κυβερνήσεις να κάνουν αυτό που πρέπει. Θα φροντίσετε το δικαίωμα πρόσβαση σε έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό να το έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ανεξαιρέτως. Η σύντομη απάντηση στην ερώτησή σας είναι ναι. Θα μπορούσα να σταματήσω και εδώ, εάν δεν πήραζε κανέναν κανένα εδώ στην αίθουσα. Διότι προφανώς αυτή είναι η υποχρέωσή μου και ο νόμος είναι νόμος. Όταν ε, κάποιος νόμος εγκρίνεται πρέπει να εφαρμόζεται. Η γενική μου λοιπόν προσέγγιση ως προς τη χάραξη νομοθεσίας και την ε, πρόβλεψη κανόνων είναι ότι εάν θέλει κανείς να έχει μια αναλογική προσέγγιση στην νομοθεσία είναι βασικά ότι όταν κάποιο νόμος ε, εγκρίνεται πρέπει και να εφαρμόζεται. Άρα θα έλεγα, εάν είχα κάποια μαγική λύση, να υπάρχουν λιγότεροι νόμοι, αλλά νόμοι ε, αυστηροί που να εφαρμόζονται αυστηρός και όχι περισσότεροι. Δηλαδή, σε κάθε τομέα αρμοδιότητας που έχω να λάβει, ένας νόμος είναι νόμος που πρέπει να εφαρμόζεται. Και ως προς αυτό που υπονοείται, πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό και ούτω καθεξής. Ένα από τα πράγματα που γενικώ θα με απασχολήσουν ε, ιδιαιτέρως και ελπίζω και εσείς και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής σας να με βοηθήσετε στην προσπάθειά μου είναι πώς την ερχόμενη πενταετία να βρούμε κι άλλους τρόπους να επιτυγχάνουμε χειροπιαστά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες και από τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Νομίζω πια με τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε να ε, αντιμετωπίσουμε είναι να γίνει κάτι το απτό για τους πολίτες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που λένε οι περισσότεροι είναι ότι δεν, μπορεί να καταλα... ότι δεν καταλαβαίνουν τι τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό αισθάνονται απομακρυσμένοι. Έτσι λοιπόν πρέπει να δείξουμε κάποια πράγματα που έχουν γίνει χειροπιαστά τα τέλη περιαγωγή, οι πτήσει ή ε, η πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Αυτά πρέπει να φανεί ότι οφείλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μας ώστε να θυμίσουμε στον καταναλωτή ποια είναι τα ωφέλη που μπορούμε να του προσφέρουμε με καλύτερα προϊόντα και σε εκατομμύρια συμπολιτών μα. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Σύρπα Πιετικάινεν από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ στην ερώτησή μου. Θα ήθελα λιγάκι να δω τι θα γίνει στο μέλλον στην Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Θα ήθελα να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των διάφορων τομέων που αφορούν την ανάπτυξη και εδώ η ερώτησή μου. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση σε σχέση με την αποδοτικότητα των πόρων αλλά και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που θα πρέπει να καλύπτονται από όλες τις πολιτικές μας προτεραιότητες και σε κάθε χάραξη πολιτικής. Πώς θα προετοιμαστείτε σχετικά ε, ω προ του δημοσιονομικού και του χρηματοπιστωτικού κανονισμού. Δεν περιμένω λεπτομέρειε σχόλια για κάθε νομοθέτημα. Αλλά θα πρέπει να να σκεφτούμε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους λόγου χάρη με την αξιολόγηση επιστοληπτικού κινδύνου και σε σχέση και με άλλα νομοθετήματα πιο συγκεκριμένα. Γενικώ ποια θα είναι η προσέγγιση σας σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι ό,τι και να πω τώρα ως απάντηση θα είναι κάτι το προσωρινό, θα είναι μια προσωρινή απάντηση. Όταν ε, προηγουμένως αναφέρθηκα στο Ταμείο για τι Μικροπρόθεσμες επενδύσει και το πώ αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε να δοχετευθούν κονδύλια λόγω χάρη σε οικοδόμηση υποδομών ή σε δράσεις ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μια άλλη κατηγορία τέτοιου είδου δραστηριοτήτων είναι μέρο τη ευρύτερη προσέγγιση που θα πρέπει να αναλάβουμε για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Ξέρετε ότι αυτό μα απασχολεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήταν ένα άλλο τομέα όπου θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα ή να προσπαθήσουμε να δώσουμε κίνητρα και να επιβραβεύουμε κάποια είδη συμπεριφοράς. Ναι, υπάρχουν τρόποι είτε με την προσφορά κινήτρων όπως διάθεση κοντιλίων ή με το να αλλάξουν οι απαιτήσει κεφαλαίων λόγου χάρη που θα επιτρέψουν την ε, κατεύθυνση κάποιων επενδύσεων σε συγκεκριμένου τομεί. Δική μου προτεραιότητα θα είναι να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε σωστά την διασωλήνωση, για να το πω έτσι, τους διάβλους μας δηλαδή, για να διοικητεύονται σωστά τα κονδύλια. Θα πρέπει να δούμε τι προτεραιότητες, κοινωνικές ή άλλες, θα, ε, θα φροντίσουμε να ε, συνδυάσουμε με κάθε δραστηριότητα. 300 δις ευρώ είναι το ποσό που αναφέρεται για αυτό το ταμείο και εμένα με ενδιαφέρει να υπάρξει και χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα προς αυτό το ταμείο. Έτσι νομίζω μπορούμε να στηρίξουμε, να αντιμετωπίσουμε μάλλον θέματα όπως αυτό που αναφέρατε και να τα διερευνήσουμε περαιτέρω. Και βεβαίως ευχαρίστω να συμπληρώσω τις απαντήσεις μου και σε μεταγενέστερο στάδιο. Ευχαριστούμε. Φάμπιο Ντεμάζη από την ΚΟΕ. Θα μιλήσω τη γλώσσα της Βασίλισσας αλλά με γερμανική προφορά. Κύριε Χίλ, Ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συναντήσατε αφότου ε, προταθήκατε από τον κύριο Γιούγκερ. Δεύτερον, αναφέρατε τον Finance Watch. Υπήρξαν εδώ κάποιες διαφωνίες ε, στο σώμα μας για την χρηματοδότηση της Finance Watch από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Τι θα κάνετε με αυτή τη χρηματοδότηση. Και τρίτον, διάβασα τις απαντήσεις σας με ιδιαίτερη προσοχή ε, ελπίζω ότι διάβασα τη σωστή ε, εκδοχή. Είπατε ότι μπορεί να υπάρξει αντιφασή μεταξύ του κανονισμού για το χρηματοπιστωτικό ιδρύματα και την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πραγματική οικονομία. Σίγουρα επηρεάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Τι θα κάνετε όμως με τη διάσωση δύο μεγάλων τραπεζών στην Ευρώπη, τι σχετικές αποφάσεις θα λάβετε και τι θα κάνετε με την ε, λανθασμένη απόδοση κονδυλίων ε, χάρη στην, ε, στον υπερβολικό όγκο συναλλαγών, εξαιτία του υπερβολικού όγκου συναλλαγών. Κοιτάξτε, στην οι Βρετανοί μοναχοί είχαν πολλές φορές γερμανική προφορά και τα αγγλικά τους δεν ήταν και τόσο καλά για πολλούς αιώνες. Τώρα για το ποιους συνάντησα εκπροσώπους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αφού του προτάθηκα. Η απάντηση είναι κανέναν. Με μία μόνο εξαίρεση. Μία μόνο εξαίρεση υπήρξε. Πήρα το τρένο για να επιστρέψω στο Λονδίνο και διάβαζα Τζόζεφ Κόνραντ για να ανακουφιστώ λίγο από το βάρος των χρηματοπιστωτικών κανόνων. Και κάτι άλλο βέβαια θα μπορούσε να με διασκεδάσει. Ε, και τέλο πάντων με πλησίασε κάποιο στο τρένο που είναι λομπίστα από πλευρά των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων. Είναι νομίζω ένα εύλογο παράδειγμα του τρόπου που συμπεριφέρονται ορισμένοι άνθρωποι. Είναι το μόνο παράδειγμα όμω που μπορώ να σκεφτώ. Ήμουν κάπου, κατά κάποιο τρόπο όμοιρο σε αυτό το τρένο. Όμω, η περιγραφή των αρμοδιοτήτων μου και αυτό ακόμη πριν προταθώ προβλέπει, και αυτούς ήθελα και να δω, είναι βουλευτές, επιτρόπους, όσους ασχολούνται με το κοινοβούλιο και με τα θεσμικά όργανα. Δεν συνείδησα λοιπόν κανέναν, απολύτως κανέναν, εξ όσων εγώ γνωρίζω, ως προς τη δεύτερη ερώτησή σας. Θα είναι το ένστικτό μου και δεν ξέρω κατά πόσο είμαι ειλικρινής για τις λεπτομέρειες της χρηματοδότησης της Finance Watch, αλλά από τις ερωτήσεις που απάντησα, ξέρω βάσει των στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης ότι έχει πολύ σημαντικό ρόλο η Finance Watch και αναγνωρίζω ότι μολονότι καταρχήν Φαίνεται περίεργο να υπάρχει δημόσια χρηματοδότηση από ένα σώμα που εκπροσωπεί τους πολίτες, ε, είναι ε, ε, αλήθεια, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε ενώσεις καταναλωτών να ανταγωνίζονται και να καλύπτουν την τεχνική πολυπλοκότητα των κανόνων που αυτές οι εταιρείε μπορούν να τους παρουσιάζουν ελπίζω, νομίζω μάλλον και αναμένω ότι αυτή η χρηματοδότηση θα ε, συνεχιστεί, γιατί πρέπει να υπάρχει και ένα αντίδοτο για το λόμπι και την άσκηση πιέσεων από τους μεγάλους οργανισμούς. Σας ευχαριστώ. Εύα Ζολή των Πρασίνων. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, δύο ερωτήσεις. Πρώτο, shadow banking. Δραστηριότητες λόγω της τεράστιας οικονομικής του ικανότητας και της περιπλοκότητας μπορούν να αποτελέσουν την αιτία της επόμενης οικονομικής κρίσης. Όμως η χώρα σας αντιτίθεται σαφώς σε ορισμένες ρυθμίσεις κλειδιά και την νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νομοθετική ρύθμιση των χρηματαγορών. Ποια είναι η δική σας θέση για τη μετατροπή των ταμείων αυτών σε αλλά μετατρέψιμα. Και ποια είναι η θέση σας για το 3-person buffer, όπως προβλέπετε αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην νομοθετική της πρόταση. Η χώρα σας αντιτίθεται κάθετα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νομοθέτηση των οροσίμων, benchmarks, και στον τομέα των ε, εμπορευσίμων αγαθών και στο ξένο συνάλλαγμα είστε διατεθειμένος να αγωνιστείτε υπέρ των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ναι ή όχι. Και προβλέπετε η ΕΣΜΑ να αναλάβει τα καθήκοντα της εποπτείας. Σας παρακαλώ. Έληξε ο χρόνος σας, λέει ο Πρόεδρος. Για το shadow banking πρώτα, Η στάση που θα πρέπει να τηρήσουμε θα πρέπει να είναι τέτοια που να επαγρυπνούμε για, την, ε, για το ενδεχόμενο να προκύψουν νέοι κίνδυνοι. Η ίδια η λέξη shadow banking σημαίνει κάτι το σκιώδες και επομένως ανεπιθύμητο. Το γεγονός είναι πάντως ότι shadow banking είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει ένα αριθμό διαφορετικών δραστηριοτήτων συλλογής χρημάτων, ας το πούμε έτσι, που ίσως θα θέλουμε και να ενθαρρύνουμε γιατί αν δεν υπάρχουν ροές χρημάτων δεν θα υπάρξει και ανάπτυξη και αν δεν υπάρχει ανάπτυξη αυτό θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα. Σε όλου αυτού του τομεί, λοιπόν και εδώ νομίζω θα συμφωνήσω μαζί σας είναι ότι πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματική νομοθεσία και να μην προσεγγίσουμε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο που να στερήσουμε το αίμα από τις ε, επενδύσεις. Τώρα για τις ειδικότερε ερωτήσεις που κάνατε, γνωρίζω το γεγονός ότι υπάρχουν, έχουν κατατεθεί προτάσεις για τα money market funds και τα πολιτικά φορτισμένα θέματα που κρύβονται από κάτω. Είμαι διατεθειμένος να τις προωθήσω τις προτάσεις αυτές και να δω πού θα φτάσουμε με αυτές. Υπάρχουν βέβαια φιλανθρωπικοί οργανισμοί και άλλοι που χρειάζονται ασφάλεια, γιατί θέλουν να πληρώνουν μισθού στο προσωπικό του στο τέλος του μήνα. Ταυτόχρονα μου εξήγησαν και ότι υπάρχει και κίνδυνοι, υπάρχουν συστημικοί κίνδυνοι από αυτά. Γι' αυτά και μιλούμε για τη ζώνη προστασία του 3%. Βέβαια χρειάζεται περισσότερη δουλειά για όλα αυτά και θα προωθήσουμε τις σχετικές προτάσεις και θα ψάξουμε να βρούμε μια μια διέξοδο που να συμφιλιώνει, λέω και πάλι, την σταθερότητα στις επενδύσεις και την αποτελεσματική νομοθεσία. Ευχαριστώ. FDD, Steven Wolf. Είναι σαφής που βρίσκεται η πίστη σας. Ορισμένοι από το Συντηρητικό Κόμμα επένεσαν τον διορισμό σας ότι δήθεν ο David Κάμερον θα υπερασπιστεί τον τομέα μας των ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Όμως στο mission letter του Juncker δεν λέει ότι πρέπει να, να καταργήσετε την υπερβολική νομοθεσία ούτε άλλα σχετικά. Τόσο πολλοί θέλουν να σας αποτρέψουν από το να έχετε οποιαδήποτε επιρροή, ώστε ακόμα και τα μπόνους των τραπεζιτών τα αφαίρεσαν από το χαρτοφυλάκιό σας. Ενώ αυτά είναι απαραίτητα για να υπάρξει χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Και κατά έναν και τον Μπρόφσκης σας λένε junior player στην ομάδα τους. Θα μπορούν να τρέψουν τις αποφάσεις σας ανά πάσα στιγμή. Όχι μόνο εκείνοι οι ε, δύο επίτροποι που ανέφερα, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος Γιούνκερ. Αυτό δεν δείχνει ότι δεν έχετε καμιά εξουσία απολύτως για να προστατεύσετε το City of London. Το γεγονός ότι όλοι καθόμαστε εδώ σήμερα με τόσο μεγάλη συμμετοχή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δείχνει ότι η Επιτροπή ΕΚΟΝ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, λαμβάνουν πολύ, σημαντικά, πολύ σοβαρά υπόψη τους τις αρμοδιότητες των Επιτρόπων. Ως αφετηρία λοιπόν, να πάρει κανείς ως αφετηρία την ιδέα ότι οι Επίτροποι δεν παίζουν κανένα σημαντικό ρόλο και ότι επομένως η παρούσα Επιτροπή δεν έχει κανένα σπουδαίο ρόλο να παίξει, δεν νομίζω ότι είναι η σωστή αφετηρία. Θέλω να πω επίσης ότι σαφώς δεν είναι καθήκον μου και προσπάθησα να το τονίσω αυτό. Εγώ δέχτηκα τον διορισμό με καλή πίστη για να προσέλθω εδώ να εργαστώ προς το γενικό συμφέρον ως Ευρωπαίος Επίτροπος. Δεν ήρθα εδώ για να προωθήσω τα συμφέροντα ιονδήποτε ομάδων. Καθήκον μου θα είναι να φροντίσω να έχουμε ένα καλά αριθμισμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πιστεύω ότι ένα καλά αριθμισμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα αποβεί προς όφελος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παντού. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει ένταση ανάμεσα στην ορθή νομοθετική ρύθμιση και στην επιτυχία του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε στέρεο κλάδο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, διότι θεωρώ ότι αν δεν έχουμε τέτοια, τέτοιες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δεν θα έχουμε ούτε τις επενδύσεις, ούτε την ανάπτυξη, ούτε την απασχόληση που χρειαζόμαστε. Αν λοιπόν θέλετε και καλά για εσωτερικούς πολιτικούς σκοπούς να μην παρουσιάσετε ψευδός ως κάποιον ο οποίος θέλει να υπερασπιστεί ένα τμήμα μονάχα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που έχει την έδρα του Λονδίνου, αυτό θα ήταν λάθος. Ευχαριστώ. Πολ Τάγκ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Τι ακριβώς σημαίνει Capital Market Union. Καταλαβαίνω πάντως ότι θέλετε να μελετήσετε περισσότερο. Να σας ρωτήσω ωστόσο κάτι το σχετικό και να εκφράσω και μια ανησυχία. Θέλετε, λέτε, να αναλάβετε πρωτοβουλία και να υποβάλλετε προτάσεις για αυτή την Capital Market Union. Αντίθετα με το ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια και να φύγετε από το ρυθμισμένο μέρος στο μη ρυθμισμένο. Δηλαδή αυτή η ένωση των κεφαλαίων να είναι ένας τρόπος απορρίθμισης περισσότερο παρά διατήρησης του ρυθμιστικού πλαισίου. Όχι, δεν το πιστεύω καθόλου. Γιατί προκειμένου να υπάρχει μια εύρυθμα λειτουργούσα έννοια αγορά, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες με τους οποίους ε, όλοι θα μπορούν να λειτουργούν. Έχουμε βάλει κάποια βασικά κομμάτια ήδη σε ό,τι αφορά το single rule book, σε ό,τι αφορά τα securities και ίσως θα πρέπει λοιπόν στον ίδιο δρόμο να κινηθούμε και να επεκτείνουμε τα ήδη. Αυτά που ήδη έχουμε κάνει. Η απάντηση στην ε, ερώτησή σας είναι ουσιαστικά ίδια με αυτή που έδωσα και προηγουμένως τον κύριο Γούλφ. Ξέρω ότι κάποιες, κάποιες φορές ή κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μια διχοτόμηση και ένα δίλημα. Είμαστε υπέρ του κανονισμού, της ρύθμισης ή υπέρ της ε, ανάπτυξης. Νομίζω ότι είναι ψευδές το δίλημα αυτό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μην υποκύψουμε στον πειρασμό, να το θεωρήσουμε δίλημα γιατί νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη είναι το πώς θα δημιουργήσουμε ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης για τους πολίτες μας. Δεν θεωρώ ότι το... είναι διαζευτικά αυτά τα δύο και αντιφατικά. Θεωρώ ότι με σωστή ρύθμιση μπορούμε να πετύχουμε ανάπτυξη. Προφανώς δεν θέλουμε υπερβολική ρύθμιση, κανείς δεν το θέλει αυτό, όλοι θέλουμε αναλογικότητα ακόμα και στην νομοθεσία. Συζητήσαμε και προηγουμένως το πώς μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ των διαφόρων ειδών επενδύσεων, πώς μπορούμε να παροτρύνουμε ε, υψηλή ποιότητα, τίτλοποίηση και πιο ασφαλή τιτλοποίηση, όπου μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις χωρίς όμως να σπρώχνουμε τον κόσμο σε πιο επικίνδυνα, σε πιο επικίνδυνα προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λαμασούρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, μία ερώτηση για την οποία ο πρόεδρος Δράγκης τόσο δεν θέλησε να μου απαντήσει. Η κρίση της τράπεζας Lehman Brothers οδήγησε τους G20 να συστήσει σε όλα τα μέλη της μία σημαντική ρύθμιση, ενίσχυση της ρύθμισης μάλλον, των τραπεζών τους κλπ. Έχουμε καμιά φορά την εντύπωση ότι με μια σαρανταριά κείμενα που είχε προτείνει ο προκάτοχός σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε ως ο καλός μαθητής των, για τι συστάσεις των G20 και ότι ωστόσο οι αμερικανικές προσπάθειες, Λότ, Φραν κλπ. ήταν είτε λιγότερο αυστηρές στα κείμενά του, είτε στην εφαρμογή του. Συμφωνείτε λίγο πολύ με την εντύπωση αυτή. Εάν ναι, η ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων παικτών υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί και αν συμβεί αυτό, αν όντω πρόκειται να συμβεί αυτό, πώς σκέπτεστε να αντιδράσετε για να το αντιμετωπίσετε. Νομίζω για να απαντήσω στην ερώτηση σας που είναι πολύ καλή ερώτηση. Πώς διασφαλίζουμε ότι οι κανονισμοί οι οποίοι ως στόχο έχουν να είναι καθολικοί και να προκύψουν από καθολικά πρότυπα εφαρμόζονται με ίσο τρόπο παντού. Η υπόθεση λοιπόν της ερώτησής σας είναι πάρα πολύ σωστή. Τώρα, για τις λεπτομέρειες, τι θα κάνω για να διασφαλίσω ότι στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα στις συζητήσεις με τις ΗΠΑ, αλλά και άλλους εταίρους, ότι υπάρχει σωστή εφαρμογή και ότι υπάρχει ε, αντιστοιχεία κτλ. Για το πώς ακριβώς θα το πετύχω αυτό, θα πρέπει να το σκεφτώ να ενημερωθώ. Αλλά για το έμεσο ζήτημα που θίγεται κατά πόσο είναι σημαντικό, ναι. Θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα, ναι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα υψηλά πρότυπα τα οποία εμείς θέσαμε τελικά δεν θα καταλήξουν να μας βάζουν σε μειονεκτική θέση σε παγκόσμιο προσκήνιο γιατί οι άλλοι καθυστερούν. Ναι. Λοιπόν, καταφατική και αυτή η απάντηση και αυτό αποτελεί ένα τμήμα της συμφωνίας TTIP. Το πώς θα πετύχουμε καλύτερη χρηματοπιστωτική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ. ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος με τον οποίο ε, μπήκαν αυτές οι διατάξεις στον πυρήνα της συμφωνίας TTIP και νομίζω ότι είναι σωστή η προσέγγιση αυτή και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα πρότυπα που συμφωνούνται από διεθνή οργανισμούς όπως η G20 τηρούνται, εφαρμόζονται και δεν βρισκόμαστε σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα γιατί εμείς τα εφαρμόζουμε και οι άλλοι δεν τα εφαρμόζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπερνάρ Μονό για τους μη εγγεγραμμένους. Κύριε Χίλ, το να οριστεί ένας Βρετανός λομπίστας που έκανε καριέρα χάρη στους ε, ιδιώτες πελάτες ή τους ε, Ρώσους ολιγάρχες είναι κάτι το παράδοξο και επίσης πώς οι κανονισμοί θα ισχύσουν στο City του Λονδίνου και θα ενοποιηθούν οι κεφαλαίοι αγορές. Οι ευρωπαϊκές αγορές, μάλλον οι ευρωπαϊκοί επίτροποι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από κάθε συμφέρον και δηλώσατε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει καμιά σύγκρουση συμφέροντος, όμως το όνομά σας συνδυάζεται με ιδιωτικά συμφέροντα όπως η υπόθεση Τέσκο. Ε, τον Ιούλιο κιόλα πωλήσατε ε, μέρος των μετοχών σας ε, για την τραπεζική βιομηχανία ε, μέρος μετοχών που, που κρατούσατε εσείς. Και όπως ο κύριος Κανιέτε, πιστεύω ότι υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος στην περίπτωσή σας. Χάρη άλλωστε, στο χρηματοπιστωτικό κόσμο τα χτίσει την περιουσία σας. Το έχει γράψει και η British Times. Πώς θα γίνει λοιπόν κύριε Χίλ ε, να αναλάβετε αυτή την αρμοδιότητα εφόσον κάνετε το πηγενέλα από την κυβέρνηση στο χώρο του λόμπι εδώ και 25 χρόνια. Πώς θα παραμείνετε ουδέτερος ε, τον ε, τομέα που έχετε αναλάβει. Ως ε, πατριώτης πρέπει να πω ότι δεν ε, προσφέρετε καμία νομιμότητα στο καθήκον που θα αναλάβετε και ότι προσωπείτε την απληστία χωρίς όρια. Παρακαλώ. Προφανώς πολύ λυπάμαι που αυτή την άποψη έχετε και η άποψη αυτή δεν προέρχεται και δεν συνάδει με την εμπειρία μου και από το πώς έχω ζήσει τη ζωή μου. Ο λόγος για τον οποίο επέστρεψα από τον ιδιωτικό τομέα, τον ιδιωτικό κλάδο στην Βρετανική κυβέρνηση, το οποίο και δεν περίμενα, είναι επειδή πιστεύω στο δημόσιο κλάδο. Ο λόγος για τον οποίο όταν μου ζήτησε ο Βρετανός Πρωθυπουργό να αποδεχτώ την υποψηφιότητά μου, πέρα από το γεγονό ότι πιστεύω ότι είναι τεράστια η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και η χώρα μου σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Ευρώπη, το οποίο είναι από μόνο του λόγος. Το έκανα όμως γιατί πιστεύω στις δημόσιες υπηρεσίες και δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφέροντων κατά οποιονδήποτε τρόπο με οτιδήποτε έκανα στην προηγούμενη ζωή μου. Όπως εξήγησα και προηγουμένως, η επιχείρηση την οποία είχα, την οποία δεν αναγνωρίζω με τα χαρακτηριστικά τα οποία της αποδίδεται, την άφησα και έφυγα πριν από πέντε περίπου χρόνια. Όσο εργαζόμουν σε αυτήν ήμουν πάρα πολύ περήφανος για τους πελάτες, για την εργασία μας. Ήμουν περήφανος που με κάποιο μικρό τρόπο και εγώ συνέδραμα στην οικονομία και στην αγορά και στην απασχόληση. Δεν αποδέχομαι την εικόνα που ε, παρουσιάζεται. Λέτε ότι είστε πατριώτης κι εγώ πατριώτη θεωρώ ότι είμαι. Είμαι βέβαιος ότι και εσεί έχετε υψηλά πρότυπα, το ίδιο και εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Μαυρίδη από τους Συνδεστές Δημοκράτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν ε, από 1,5 περίπου έτος, κάτι ανήκωστο έγινε στην τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κούρεμα των καταθέσεων, αλλά και σε όλο το υπόλοιπο θέμα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά της αρρωγής, ε, καταπήγουσας αρρωγής από μία τράπεζα σε μία άλλη, από μία τράπεζα σε πτώχευση σε μία άλλη. Και τώρα βλέπουμε ότι τα πράγματα συστημικά έχουν καταρρεύσει. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη πλέον στον τραπεζικό κλάδο που εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ αδύναμος. Και από την άλλη υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος σε ό,τι αφορά την ε, διάσωση του τραπεζικού συστήματος. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Καταρχά. Το πείραμα της Κύπρου έχει στεφθεί με επιτυχία τελικά. Και ποια είναι τα διδάγματα από τα παθήματα της Κύπρου σε περίπτωση που παρουσιάστηκε μια ανάλογη περίπτωση. Κατά δεύτερον, είπατε και ότι είσαστε ρεαλιστής και πραγματιστής. Πιστεύετε πραγματικά ότι στην περίπτωση της Κύπρου, έχοντας υπόψη την περίπτωση της Κύπρου, θα υπάρξει ε, μια τραπεζική ένωση χωρίς ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο για τις καταθέσεις. Απάντηση. Κατανοώ προφανώς τις ιδιαίτερα δύσκολες περιστάσεις ε, και δυσκολίες που αντιμετώπισε η Κύπρος. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην ε, συμπονούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Ρωτάτε αν μάθαμε από το παθήματα, από τα μέτρα που ελήφθησαν για να εισαχθεί ένα σχέδιο εγγύησης καταθέσεων προκειμένου στο μέλλον, σε περίπτωση που θα προέκυπτε μία παρόμοια κατάσταση, θα υπήρχε μία εγγύηση για 100.000 καταθέσεις. Αυτή είναι η απάντηση νομίζω για το πώς θα κινηθούμε στο μέλλον. Τώρα, για το κατά πόσον θα υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για τις εγγύησεις καταθέσεων, το συζητήσαμε λίγο πριν αυτό το θέμα. Ξέρω ότι υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ, υπάρχουν επιχειρήματα κατά ενό τέτοιου σχεδίου. το να προχωρήσουμε το σχέδιο που ήδη υφίσταται και έχει εφαρμοστεί σήμερα είναι ο σωστός τρόπος, θεωρώ, για το μέλλον. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια ενδιάμεση αναθεώρηση, αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Ευχαριστούμε. Από το ΕΛΚ, Brian Hayes. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να καλωσορίσω τον Λόρδο Χιλ αυτή την ακρόαση. Πρώτα απ' όλα για τις κεφαλαίες Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, χρειάστηκε μια ολόκληρη οικονομική κρίση για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, να δημιουργηθεί η Τραπεζική Ένωση. Και όπως είπε βέβαια και ο συνάδελφος, πολλά απομένει ακόμη να υλοποιηθούν. Πώς θα υπάρξει ένωση κεφαλαίου αγορών στο μέλλον. Πώς βλέπετε το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για να υπάρξει μια τέτοια ένωση. Και τι στόχους θα περιμέναμε από την ένωση των ε, κεφαλαγορών. Το backlanding πώς θα το ε, ενθαρρύνουμε ε, ή πώς θα το εμποδίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν είμαι υπέρ θα πρέπει επίσης να δούμε τα ωφέλη της ενίας αγοράς για τους ε, πολίτες, όπως τις ε, ψηφιακές πληρωμές που αναφέρατε. Στην Επιτροπή μας μπορείτε να πείτε τι προτάσεις θα υποβάλλετε για να υπάρξει σωστή διευθέτηση των ψηφιακών νομισμάτων. Ε, μία από τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται, αλλά που θα μπορούσε να εξελιχθεί και σε απειλή. Ευχαριστώ για αυτές τις δύο ερωτήσεις. Ξέρω ότι δουλειά έχει γίνει και στο παρελθόν με την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών. Εκεί προβλέφθηκε μια σειρά από μέτρα για τις επιγραμμικές πληρωμές, ιδίως οι σωστές πληροφορίες για τους πελάτες, χωρίς να υπάρχει δηλαδή κίνδυνος ασφάλειας με τις κατάλληλες υπηρεσίες. Για άλλα ψηφιακά ε, νομίσματα όπως το bitcoin αυτά νομίζω ότι απασχολούν πολύ τις ε, συζητήσεις μας και πρέπει να βρεθεί το σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ κινδύνου και καινοτομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, τις, για τα ψηφιακά νομίσματα ε, πήρε μέρος σε μια ακρόαση που η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και θα υπάρξουν και τριμερείς διάλογοι, θα συζητηθεί δηλαδή και αυτό το θέμα εκεί, στα πλαίσια της οδηγίας ε, για την ελεύθερη παράνομων προσόδων. Θα το παρακολουθούμε λοιπόν αυτό με ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα ως προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών θα χρειαστεί άλλη κρίση ενδεχομένως. Νομίζω πως όχι. Αυτό τουλάχιστον ελπίζω και δεν θα έπρεπε να το δούμε το θέμα έτσι. Έτσι χρειάστηκε να προσεγγίσουμε και το θέμα της Τραπεζικής Ένωσης. Ελπίζουμε ότι το τοπίο θα είναι κάπως πιο ε, ήρεμο και ως προς το χρονοδιάγραμμα νομίζω ότι Πρώτα θα πρέπει να αναλύσω και να εξετάσω προσεκτικά τα θέματα σε διαβούλευση και με άλλους και ως προς το backstop που σας ανέφερα, τον ανασταλτικό μηχανισμό. Στην επιστολή αρμοδιοτήτων που έλαβα είναι πολύ σαφές ότι αυτό θα πρέπει να λειτουργεί πλήρως μέχρι το 2019. Εγώ νομίζω ότι στοιχεία θα παρουσιαστούν ε, ήδη στο άμεσο μέλλον προκειμένου να έχουμε λόγω χάρη υψηλής ποιότητας τυλοποίηση πολύ πιο γρήγορα. Αυτό πιστεύω θα συμβεί στο άμεσο μέλλον μέλλον, ίσως και στις αρχές του επόμενου χρόνου. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. σαν ποτέρχο από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στο ότι το αυξημένο επίπεδο τραπεζικών κανονισμών δημιουργεί σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, υπάρχει ένα πραγματικό κίνδυνο να προτείνεται υπερβολικά πολλή νομοθεσία. Λόγου χάρη, νωρίτερα φέτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό για τι τράπεζε και τι διαφορετικέ του μεταρρυθμίσει που δεν θα επιτρέπουν στι τράπεζε να έχουν ξεχωριστές αγορές ε, για συγκεκριμένα παράγωγα προϊόντα τους. Υπήρχαν λοιπόν διορθωτικοί περιορισμοί που ενδεχομένως όμως να είναι βλαβεροί για τους ε, πελάτες των τραπεζών. Δεν θα μπορέσουν να παράσχουν υπηρεσίες ή τίτλους ή τράπεζε βάσει τη παλιά του χρηματοδότηση. Θα φροντίσετε εσεί να προβλεφθεί τέτοια νομοθεσία ώστε οι εταιρείε να έχουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Και πώ θα το διασφαλίσετε, πώ θα μπορέσει η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών να τροφοδοτείται από διαφορετικέ πηγέ χρηματοδότηση και πώ επίση θα ωφελήσει τι μικρομεσαίες επιχειρήσει χωρί να είναι ε, ένα, ένα στοιχείο περιορισμού και μόνον. Μάλιστα. Πολύ πιστό στο χρόνο σας. Το βασικό σας επιχείρημα για την σωστή προσέγγιση ως προς την ε, νομοθεσία και πώς δεν θα έχουμε υπερβολικά πολλή νομοθεσία. Παραλείποντας κινδύνους που αναδύονται ή προκύπτουν. Αυτή είναι μια πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε όλοι μας, και εγώ και οι άλλοι στην εξάσκηση των καθηκόντων μας. Δεν είναι απλό ούτε λογικό να δώσω μια απλή απάντηση στο τι θα κάνω. Σίγουρα πρέπει κανείς να κρίνει αναπερίπτωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό βεβαίως διαρκώς να το ελέγχει για να είναι βέβαιος ότι η απόφαση ήταν σωστή. Διότι αν δούμε το τεράστιο όγκο νομοθεσία και επιτευμάτων μα τα τελευταία πέντε χρόνια, νομίζω με την κοινή λογική μπορούμε να πούμε ότι αν νομοθετούμε με τέτοια ταχύτητα και υπό τέτοια πίεση, προφανώ δεν μπορεί όλα να ήταν σωστά ε, και εύστοχα ευθύ εξ αρχή. Νομίζω λοιπόν η προσέγγιση του κοινού νου είναι να βλέπουμε τα πράγματα ξανά διαρκώ και διαρκώ για να προσαρμόζουμε. Μερικέ αναθεωρήσει προβλέπονται ήδη εντό τη νομοθεσία. Νομίζω εκατοντάδε τέτοιε αναθεωρήσει προβλέπονται τα επόμενα πέντε χρόνια που θα πρέπει να ξαναδούμε τον αντίκτυπο τη νομοθεσία. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά εάν θέλουμε μια συνεκτική ε, θεώρηση ολόκληρη τη νομοθεσία και ω προ τη διεθνική μεταρρύθμιση και τις προτάσεις Λικάινεν, οι προτάσεις του Αντιπροέδρου Μπαρνιέ ε, για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της εξάλληψης κινδύνου που δεν θα πλήττει το ενιαίο τραπεζικό ε, μοντέλο, την ε, εμπορία τίτλων ιδιοκτησίας. Αυτό ε, νομίζω κατά την άποψη κάποιων είναι υπερβολικό, κατά την άποψη κάποιων άλλων όχι. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να προωθήσουμε την όλη πρόταση, να δούμε που θα φτάσουμε και να αναζητήσουμε την κατάλληλη ισορροπία. Ευχαριστούμε κύριος Γέντζεκ για, την, για τους φιλελευθέρους. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, θα ήθελα να επανέλθω στο ζήτημα των money market funds και το 3% ζώνη προστασίας. Μπορεί κανείς να συναγάγει από τις απαντήσεις σας ότι προτίθεστε να επανεξετάσετε την πρόταση που έχει υποβάλει στη διαδικασία ο προκάτοχός σας. Μου μένουν λίγα δευτερόλεπτα. Να επανέλθω στις κεφαλαιαγορές. Πού εντοπίζονται εμπόδια στην ενιαία αγορά και προτίθεστε να ολοκληρώσετε την ενιαία αγορά με οδηγίες ή με κανονισμούς. Απάντηση του Λόρδου Χιλ για τα money market funds πρόθεση δική μου θα είναι μάλλον να προχωρήσουμε με την πρόταση ή με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί ήδη, όπως έλεγα πριν. Αυτή θα είναι η προσέγγιση μου. Συνήθως συνεχίζεται η διαδικασία συζητήσεων. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αποσύρθουν οι προτάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να τις εξετάζουμε και όσον αφορά την ΣΥΝΑΦ ή τη ΣΥΝΑΦΣ νομίζω πρέπει να ψάξουμε να βρούμε μια λύση που να επιτρέψει σε αυτά τα ταμεία να διατηρούν το ρόλο τους μέσα στην οικονομία ταυτόχρονα διασφαλίζοντας την οικονομική σταθερότητα. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση για την ένωση των κεφάλαιων αγορών. Κατανοώ την επιθυμία να ακούσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά όπως είπα και πριν, νομίζω ότι πρέπει να τις αναπτύξουμε, ε, να προχωρήσουμε βήμα-βήμα, να δούμε δηλαδή πρώτα προς τα πού θα πρέπει να προχωρήσουμε. Και αν τώρα θα ενδυθούν το ένδυμα του κανονισμού της οδηγίας, ακόμα δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση γι' αυτό. Όταν θα έχει διαξαχθεί ανάλυση και θα έχουν τα προβλήματα, τότε θα δούμε ποια βήματα θεωρούμε ότι πρέπει να λάβουμε για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά ή να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να μπορεί να κινηθούν, να ρεύσουν τα κεφάλαια και ιδίως προς αυτούς που τα έχουν ανάγκη, είτε για επιχειρήσεις είτε για άλλους σκοπούς. Ζαντ, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Χώρες μέλη και περιφέρειες. Έχουν εκεί ορισμένα πλεονεκτήματα ανταγωνισμού. Ορισμένες περιφέρειες, ωστόσο, έχουν αναπτύξει μια αρμοδιότητα για την παραχώρηση για την χορήγηση μάλλον ε, υπηρεσιών κοινή ωφέλεια, όπω Κύπρο, ε, ε, Γιβραλτάρ κλπ. Οι financial services μπορούν να προωθήσουν ωστόσο την ένταξη στην αγορά. Το ίδιο οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μπορούν να προωθήσουν την οικονομική δραστηριότητα και τις δουλειές σε ορισμένες περιφέρειες που αλλιώς είναι καταδικασμένες σε μια στασιμότητα. Αυτά τα στάνταρ τα προδιαγράφει ο ΟΣΑ. Θεωρείται ότι η παροχή τέτοιων υπηρεσιών από περιφέρειες θα πρέπει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί. Το βασικό νομίζω που πρέπει να επιδιώξουμε είναι να φροντίσουμε ότι οι υπηρεσίες προσφέρονται από οποιονδήποτε ότι αυτές προσφέρονται σε πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού. Δεν μπορούμε να δεχθούμε κάποιοι να δρούν υπό κανόνες ελαφρότερους από άλλους. Ο... Η αρχή που πρέπει να υιοθετηθεί είναι να διασφαλιστεί ότι συνολικά, όπου και αν βρίσκεται κάποια περιφέρεια, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μέσα σε πλαίσιο ίσων όρων ανταγωνισμού. Και επομένω χρειάζεται διαφάνεια, είτε θεσπισμένη από τον ΩΣΑ είτε από, άλλα, από άλλους οργανισμούς. Και αυτά, τα, αυτές τις προδιαγραφές πρέπει να τις διατηρήσουμε. Ευχαριστούμε. Φλάβιο Μαρτουσέλο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Επίτροπε, δεν ξέρω αν διαβάσατε χθες τη δήλωση του ε, Πρόεδρου της ε, Τραπεζικής Ένωσης που λέει ότι είναι πολλές οι τράπεζες που σύντομα πρόκειται να πτωχεύσουν. Ή τέλος πάντων είναι κάποιες τράπεζες που πρόκειται να πτωχεύσουν άμεσα. Είναι χρήσιμες τέτοιες δηλώσεις από την άποψη του χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Και εσείς πώς θα τις αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους δηλώσεις. Επίσης χθες το κράτος της Ιταλίας δήλωσε ότι η υποβολή σχεδίου προπολογισμού αναβάλλεται. Ε, το ίδιο έκανε και το Βέλγιο για τη συμμόρφωση ε, με τους στόχους ε, του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν θα υπάρξουν επιπτώσεις μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες από τέτοιου είδους εξελίξεις. Ευχαριστώ Δεν νομίζω ότι ε, έλαβα γνώση των συγκεκριμένων σχολείων που αναφέρατε. Ως... Με συγχωρείτε, είμαι κάπως ε, ε, βραδύς ίσως και δεν κατάλαβα την ερώτηση που υπονοείται για την Τραπεζική Ένωση. Μπορείτε... Να μου πείτε τι ακριβώς ρωτήσατε. Χθε στη Βιέννη, ο Αντρέ Δία, κάτι που το μετέδωσαν όλα τα πρακτορία, δήλωσε ότι κάποιες τράπεζες δεν θα περάσουν τον έλεγχο κόποση, τον έλεγχο αντοχή και θα πτωχεύσουν. Με τέτοιου είδους δηλώσει. πώς θα κεφαλοποιείτε το σύστημα και εσείς θα κάνατε στη θέση του κυριορία τέτοια δήλωση. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Δεν ε, κατάλαβα ότι είπατε για έλεγχο κόπωσης. Δεν μπορώ να προδικάσω τα αποτελέσματα του ε, ελέγχου κόπωσης, αντοχής μάλλον, ε, συνεχίζεται και τα αποτελέσματα τα αναμένουμε. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της όλης διαδικασίας ε, του να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ισχυρές και σταθερές τράπεζες στην Τραπεζική Ένωση. Γνωρίζω ότι οι τράπεζες έχουν λάβει μέτρα για να αυξήσουν το κεφάλαιό τους. Ξέρω ότι η διαδικασία αυτή είναι κάτι που έχει απασχολήσει όλους σοβαρά και με αυστηρότητα, με πολλή πειθαρχία. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε τα αποτελέσματα του ελέγχου όταν ολοκληρωθεί, αλλά σε αυτή τη φάση δεν το βρίσκονται λογικό ούτε συνετό να σχολιάσω το τι θα μπορούσε να συμβεί. Διότι δεν ξέρω τι θα πούν. Όμως το να ισχύει αυτό το τμήμα της υποδομής που χρειαζόμαστε ώστε να γνωρίζουμε βάσει της λογικής με ποια βάση θα προχωρήσουμε με την Τραπεζική Ένωση βρίσκω ότι είναι το σωστό. Και τα αποτελέσματα θα τα ξέρουμε σύντομα. Ελπίζω το νέο σύστημα που θα ισχύσει για το μέλλον με το Συμβούλιο Εξυγίανσης, το Ταμείο Εξυγίανσης και ούτω καθεξής θα προσπίσει καλύτερα τα συμφέροντά μας και στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μαλέτιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κύριε Υποψήφιο Επίτροπε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι με, έχει να κάνει με τα υψηλά επίπεδα δανειοδότησης και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Τι θα γίνει σε περίπτωση που υπάρξει αποτυχία στις επιχειρήσεις και αφαιρεγγιότητα για το insolvency, πώς θα λειτουργήσει η νομοθεσία και στην όλη διαδικασία στηρίξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ο κανονισμός για τις πληρωμές. Τι άποψη έχετε για τον κανονισμό των πληρωμών. Και τι πιστεύετε για τις πληρωμές στα κρατη Θα πρέπει να γίνονται οι πληρωμές προς τους ε, πιστωτές μέσα σε 60 ή 90 ημέρες το πολύ. Από την άλλη αντιμετωπίζουμε δυσκολίες με πληρωμές από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό προς τα κρατη Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επιλύσουμε το ζήτημα αυτό. Εσείς τι θα κάνετε σχετικά. Νομίζω πολλά από αυτά είναι θέματα που δεν άπτονται στην, της καρδιάς του χαρτοφυλακίου μου, για να το πω έτσι. Όμως, θα είμαι μέλος του Σώματος των Επιτρόπων που εξετάζει αυτά τα θέματα. Βεβαίως γνωρίζω τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν επιχείρηση συστάσεις και σε σχέση με τη σταθερότητα που επιδιώκουμε, όμως αυτό είναι μια αρμοδιότητα κατεξοχήν του κυρίου Μοσκοβισή, ο οποίο θα πρέπει με του δικού του συνεργάτε να το δει. Ω προ τα επίπεδα των πληρωμών, ναι, γνωρίζω ότι έχουν ληφθεί κάποια πρώτα μέτρα ω βήματα για την οδηγία των πληρωμών, ένα ξεχωριστό θέμα. Όμω, εάν μετά από αυτήν την συνάντηση μπορέσουμε κάποια ζητήματα να τα δούμε διμερώς και να μου εξηγήσετε τις ειδικές σας ανησυχίες, ευχαρίστω θα το πράξω. Ευχαριστούμε. Γιώνας Φερνάντεφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Χίλ. Θα μιλήσω τη γλώσσα του Φερβάντες. Ο κύριος, ο κύριος Μπαρνιέ ήταν ιδιαίτερα δραστήριος ε, κατά την προηγούμενη θητεία ώστε να εξετάσει τουλάχιστον 50 νομοθετικές προτάσεις η Επιτροπή μας που άπτονταν των αρμοδιοτήτων του. Κάποιες από αυτές ε, έγιναν πολύ ποιότερες χάρη στην νομοθετική μας εργασία. Εσείς θα είσαστε το ίδιο δραστήριο με τον κύριο Μπαρνιέ ή θα είσαστε πιο πραγματιστής και θα είσαστε λιγότερο φιλόδοξος από ό,τι στην αρχή της θητείας. Ε, έπειτα θα γνωρίζετε ότι η ε, Επιτροπή μας ασχολείται με το θέμα των ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Υπάρχουν πιέσεις για να ε, για να αλλάξει ο ορισμός του κάθε δίκτυ, ο οποίος να μπορεί να ελεγχθεί και να υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία ε, παρακολούθησης. Πιστεύετε ότι το θέμα των δικτών μπορεί να ξανανοίξει ή μπορεί αναδείκτη να έχουμε μια απορρίθμιση ανάλογα με τη σημασία τους. Αυτό βεβαίω θα ανοίξει τη βασιλική οδό για τη δημιουργία περαιτέρω γραφειοκρατία. Ελπίζω ότι και αν κάνω να μην ε, στραφώ κατά των ανεμομήλων κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως προς την ε, ε, νομοθεσία και την ποσότητά της θα ακολουθήσω το παράδειγμα του κ. Μπαρνιέ προφανώς αλλά πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής ότι επειδή ήταν μεγάλος όγκος της νομοθεσίας που πέρασε τα τελευταία χρόνια Πρώτη μου προτεραιότητα είναι 400 περίπου μέτρα που μαζί μας θα πρέπει, μεταξύ μας μόνο θα πρέπει και να τα εξετάσουμε και να τα εγκρίνουμε και να τα υλοποιήσουμε. Η πρώτη μου λοιπόν απάντηση είναι ότι θα υπάρξει πολλή δουλειά επί των λεπτομεριών και θα είμαστε ιδιαίτερα απασχολημένοι. Επίσης γνωρίζουμε ήδη ότι κάποια πράγματα που έχουμε συζητήσει εκεί για τα money market funds, για τη συγκεντρική αξιολόγηση, μπορεί να χρειαστεί και άλλη δουλειά. Κάποια διευθυντικά θέματα που αφορούν τις τράπεζες, οι αναδυόμενοι κίνδυνοι, ή για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών να χρειαστεί ενισχυτική συμπληρωματική νομοθεσία. Αλλά για την ερώτηση που υπονοείται μέσα από όσα είπατε. Εάν θα μπορέσουμε να βρούμε με αυτό το δύσκολο και άπιαστο σημείο ισορροπίας μεταξύ του μεγάλου όγκου νομοθεσίας ώστε το σύστημα να είναι ασφαλές αλλά όχι τόσο ασφαλές που να εμποδίζει την, ε, τις οικονομικές συναλλαγές και δραστηριότητε. Δεν μπορώ λοιπόν να σας δώσω μια απάντηση σε αριθμούς δεν έχω να σας πω κάτι σε ποσοστό ή σε μέγιστο ανώτατο όριο, διότι και ο κύριος Μπαρνιέ ο ίδιος είχε πει ότι θα νομοθετήσει όσο χρειαστεί, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που παρουσιάζονταν. Αυτή είναι και η δική μου προσέγγιση. Νομίζω το μόνο που θα είχα να προσθέσω είναι ότι θα έπρεπε να δούμε τι κάναμε στο παρελθόν, να βεβαιωθούμε ότι τα κάναμε σωστά και ξέρω ότι σε αυτό θα συμφωνούσε και ο κύριος Μπαρνιέ. Για τα benchmark στην συγκριτική εξολόγηση θα πρέπει να απαντήσω στα πλαίσια άλλης ερώτησης. Κυρία Ματίας από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ. Κύριε Χίλ, Όπως ξεκινήσαμε τη γλώσσα αυτή, την συζήτηση αυτή, θα μιλήσω και εγώ τη γλώσσα του Καμόης και του Σαραμάγκου. Ήδη είχα την ευκαιρία να το συζητήσω αυτό προσωπικά μαζί σας. Όταν προέκυψε η οικονομική κρίση, αυτό που δεν έλειψε ήταν υποσχέσεις που έλεγαν ότι θα διευθετηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είπατε προσωπικά και το συμμερίζομαι και εγώ ότι προσποιήθηκαν ότι τακτοποιούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα ή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν έγιναν λοιπόν πολλά και γι' αυτό έχω συγκεκριμένε ερωτήσεις. Πρώτον, για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μίλησε για την έκπτωση φτηνού χρήματο που θα διοχετευτεί στην οικονομία η Κεντρική Τράπεζα. Όμω αυτή η ρευστότητα δεν θα επηρεάσει τι πολιτικέ επενδύσεων που επηρεάζουν με τη σειρά του την οικονομία. Η έλλειψη ρευστότητα δεν μας προετοιμάζουν για, για την επόμενη χρηματοπιστωτική κατάρρευση. Έπειτα για την θεσμική διάρθρωση των τραπεζών θα προχωρήσετε για, την, για τη διευθέτηση αυτού του θέματος. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. 20 δευτερόλεπτα. Η τρίτη ερώτηση είναι αν μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση που έθεσε ο συνάδελφος για, τους, ε, ε, υπόγειους, ε, για την υπόγεια χρηματοδότηση που δίνεται στις αποτυχημένες, τις, κατεστραμε, τις πτωχευμένες τράπεζες. Κατά πρώτον, για το κατά πόσον όλη η δουλειά του προκατόχου μου την τελευταία πενταετία δεν είχε σοβαρό αντίτυπο ε, και κατά πόσον ήταν ε, πεταμένος, χαμένος χρόνος. Νομίζω ότι όλοι θα συμμεριστείτε σε αυτή την Επιτροπή την άποψη που θα εκφράσω χρειάστηκε να βρεθούν απαντήσεις υπό συνθήκες πίεσης, έκτακτες συνθήκες. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε την κατάρρευση του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, του τραπεζικού μας συστήματος και όλων των υποδομών που διέπουν τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Τώρα, κάτι διασώσαμε, γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ και αυτό είναι ένας φόρος τιμής που πρέπει να αποτίσουμε. Τους διασώστες Ξέρω ότι είσαστε από αυτού που θα θέλατε να έχουν γίνει και περισσότερα. Όμω, προκειμένου να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπία και να αναλάβουμε την ε, απαραίτητη δράση ώστε να υπάρξει σταθερότητα στο σύστημα, νομίζω και ο προκατοχό μου και το σώμα σα έχουν λόγου να πιστεύουν ότι πέτυχαν σωστά αποτελέσματα. Ως προς την Κεντρική Τράπεζα και τα ιδιωτικά κονδύλια το ιδιωτικό χρήμα, μέρος της αρμοδιότητάς μου, και ελπίζω να το πετύχω αυτό με την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών, είναι να εξεύρω τρόπους ώστε τα κονδύλια από, την, από τον ιδιωτικό τομέα να απελευθερωθούν και να συνοδεύσουν τα δημόσια. Η δέσμευση του κ. Γιούνκια για 300 δις ευρώ είναι μια δέσμευση που θα πρέπει να βρούμε τρόπο να την μοχλεύσουμε με χρήμα του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος να έρθει και να ενωθεί με το δημόσιο και να προσπαθήσουμε έτσι να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι δεν έχω άλλο χρόνο. Για την άλλη σας ερώτηση, ίσως με, κάποια, με αφορμή κάποια άλλη. Ευχαριστώ. Τους πράσινους ο κύριος Λάμπερτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χίλ. Καλώς ορίσατε και πάλι. Ε, συναντηθήκαμε άλλη μια φορά σήμερα και είπατε κάτι που μου έκανε εντύπωση. Είπατε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπερβολικά μεγάλα ώστε να μην μπορούν να αποτύχουν. Είχατε δίκιο σε ό,τι αφορά την εκ νέου ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Έχετε δίκιο γιατί εξακολουθούμε να έχουμε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δεν μπορούμε να τις επιτρέψουμε να φαλυρίσουν. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ. Έχω να ρωτήσω το εξή. Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά μέτρα τα οποία θα θέλετε να πάρετε για να διασφαλίσετε προκειμένου να μην υπάρχουν όντως, όπως είπατε, ιδρύματα υπερβολικά μεγάλα για να αποτύχουν για να μπορούμε να τα διχειριστούμε και ούτω καθεξής. Απάντηση. Νομίζω ότι είναι σημαντική η ερώτηση αυτή και έχουμε συνδεθεί και άλλες φορές, όχι μόνο μία φορά. Ποιοι είναι οι άλλοι κίνδυνοι Δεν ξέρω ποια είναι η προσωπική σας άποψη, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να θέσουμε σε εαυτούς μας την πρόκληση του να αντιμετωπίσουμε τα ιδρύματα τα οποία είναι υπερβολικά μεγάλα ε, και δεν μπορούμε να τα εξηγιάνουμε, δεν μπορούμε να τα διαλύσουμε. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Καταρχάς, θα πρέπει να σταματήσουμε το πρόβλημα προτού εμφανιστεί σε πρώτη φάση. Αυτό είναι ένα τμήμα της συζήτησης που θα γίνει για τις διαχρητικές μεταρρυθμίσεις. Το ξέρω. Θα προσπαθήσουμε να άρουμε τον κίνδυνο από αυτή την πλευρά της πρόκλησης. Θα πρέπει γενικά να επιμείνουμε στη λογική του γνωρίζουμε που έγινε ο κίνδυνος στο θέμα της διαφάνειας το θέμα στο ότι σε μια σειρά χρηματοπιστωτικών ενδερμάτων, όχι μόνο στις τράπεζες, θα είμαστε, θα έχουμε συνείδηση των κινδύνων και που κρύβονται, να υπάρχουν μηχανισμοί εξυγίανση εκεί όπου τους χρειαζόμαστε και έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό κλάδο. Υπάρχουν και άλλοι κλάδοι, ξέρω, που θα ήθελε πολλοί κόσμος να πραγματευτούμε. Νομίζω ότι προχωράμε. Εγώ θα είχα ανοιχτό πνεύμα για τα μέτρα τα οποία ενδεχομένω θα, θα, θα χρειαζόταν να πάρουμε. Θα ήθελα να πάυσει αυτή η ανισότητα αυτή η αντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ νομοθεσίας και κάποιων επιχειρήσεων που είναι μεγαλύτερες από το ΑΕΠ ολόκληρων χωρών, προκειμένου να γίνουν όλα αυτά με σωστό και λογικό τρόπο. Ευχαριστώ για το, e για το ΑΕΛΚ, ο κύριος Λάγκε. Σας ευχαριστώ. Λόρτα Χίλ, στο mission letter σας αναφέρετε ότι είστε υπεύθυνο και για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Το είπατε κι εσείς. Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις του Προέδρου της Κομισιόν για τα Ευρωομόλογα, πώς τις αξιολογείτε, πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, ποια αξία θεωρείτε ότι υπάρχει στο εμπόριο υψηλής συχνότητας στα μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Και τρίτη ερώτηση, ποια σημασία έχουν για σας στο μέλλον οι πράξεις κατά αξιοδότηση. Πώς θέλετε να εμπλέξετε το Κοινοβούλιο εγκαίρως και τα τρία θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα, η Επιτροπή της Βασιλείας, η οποία στο παρελθόν πάντα αξιολογούσε μηδενικό τον κίνδυνο των κρατικών ομολόγων, αλλά αξιολογούσα τα, τις ιατρικές σχέσεις με υψηλό κίνδυνο. Πότε λοιπόν θέλετε να προτείνετε αξιολόγηση των τριών αυτών ζητημάτων τους επόμενους μήνες. Πολλές ερωτήσει πολλές ερωτήσεις μου, μου θέσατε. Κάποιες αρκετά τεχνικής φύσεως. Το λογικό λοιπόν θα ήταν να σας συναντήσω με τους ε, υπαλλήλου των μελλοντικών μου υπηρεσιών, ελπίζω, προκειμένου να το συζητήσουμε σε βάθος σε ό,τι αφορά τη γενικότερη προσέγγιση που θα υιοθετούσα για τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση και τις πράξεις της εφαρμοστικές. Θα ακολουθούσα την μέθοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό, θεωρώ, να συζητιούνται αυτά έκτενος, να γνωρίζει ο κόσμος τα θέματα και τις προτάσεις επιτάπητος και θα ήθελα αυτή τη λογική να ακολουθήσω σε όλους τους τομείς. Για τα ευρωομόλογα. Σε ό,τι αφορά τα ευρωομόλογα. Δεν είναι ιδιαίτερα ενημερημένο η απόψή μου προκειμένου να σας απαντήσω για το συγκεκριμένο αυτό το θέμα στην παρούσα φάση. Προφανώς είναι κάτι στο οποίο θα εμβαθύνω και είναι δεδεθμένος να συζητήσω μαζί σας. Thank you. And now for the e again. Η e FDD e τώρα, ο κύριος... τώρα κύριος Στέφαν Γουλφ. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί είσαστε εδώ και ποιος είναι ο σκοπός του διορισμού σας. Κάτι είπατε σήμερα ότι θα δουλέψετε προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι υπέρ κάποιων ομάδων ή χωρών. Σίγουρα αυτά θα ενθουσιάσουν τσο τους αντίθετους του David Cameron. Είπατε ότι θα εφαρμόσετε τους κανονισμούς. Είπατε ότι η Capital Markets Union θα αρχίσει ανεξάρτητα από εκείνους που δεν γνωρίζουν καν περί τίνος πρόκειται. Όμως νομίζω ότι υπάρχει και ένας άλλος στόχος για την έλευση σας εδώ. Στη σελίδα 5 της Mission Letter που ο Jean-Claude Juncker σας λέει. Θα πρέπει να βρείτε τρόπο να καταργήσετε τις, συνεισφορές των, τις δημοσιονομικές εισφορές στους τρεις ρυθμιστές που θα πρέπει να καταβάλλονται από τους εποπτευόμενους τομείς. Το Συντηρητικό Κόμμα ψήφισε πριν από λίγες εβδομάδες στην παρούσα Επιτροπή ακριβώς τέτοια έκθεση που σημαίνει στην ουσία φορολόγηση από την πίσω πόρτα της ε, του Λονδίνου. Ο διορισμός σας είναι business as usual για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Ενωμένο Βασίλειο. Απάντηση του Λόρδου Χίλ. Δεν νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω τίποτε περισσότερο στις απαντήσεις που σας έδωσα προηγουμένως. Δεν νομίζω ότι όντω αυτή είναι η δουλειά που ελπίζω ότι θα μπορέσω να εκτελέσω εδώ ως μέλος του Συλλογικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα καθήκοντά μου που ελπίζω ότι θα μπορέσω να ασκήσω εκεί θα είναι να έχουμε μια, ένα ισχυρό κλάδο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που να ωφελήσουν όλους όσοι εξαρτώνται από αυτά. Και αν έχετε μια ισχυρή τέτοια ένωση αυτή ανοίγει πολλές ευκαιρίες στους τομείς αυτούς για να αυξήσουν τις αγορές τους και να οδηγήσουν σε ανάπτυξη της επιχειρήσης τους. Είχα την εντύπωση ότι αυτό θα ε, σας ενδιέφερε γιατί γνωρίζω το ιστορικό σας στο ΣΥΡΙ του Λονδίνου. Πέραν από αυτό όμως δεν μπορώ να προσθέσω τίποτε άλλο γιατί δεν νομίζω ότι πραγματικά σας ενδιαφέρει η απάντηση που σας δίνω. Thank Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, εμείς μιλούμε για διατήρηση της πραγματικής οικονομίας και η δυνατότητα να κάνουν οι άνθρωποι και κάποιες αποταμιεύσεις. Επ' αυτού θέλω να γνωρίζω τι πιστεύει για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για να υπάρξει κάποια σταθερότητα και να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία. Αυτά τα έχει προωθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνείτε? Και δεύτερον, αν και δεν εξαρτάται απολύτως από εσά. Θα, συμφων... θα συμμετάσχετε ωστόσο για τη φορολογική βάση και για το συντελεστή αυτού του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και τρίτο, δεν έχω καταλάβει πολύ καλά την απάντησή σας στην κυρία Περβάν Σουμπερές για την οδηγία για το πλήσιμο του βρώμικου χρήματος. Σας έχει αφαιρεθεί αυτό, που νομίζω ωστόσο ότι είναι ένα ρυθμιστικό εργαλείο το οποίο θα σας λείψει δεν κατάλαβα πολύ καλά και την απάντησή σας. On the... Uh, Ο Λόρδος Χιλ. Πρώτα για τον φόρο, FTT. Θέμα που όπως γνωρίζετε είναι της αρμοδιότητας του κ. Μοσκοβισή. Ο πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε ότι γι' αυτόν η φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι ζήτημα ε, δικαιοσύνης. Έχει γίνει η πρώτη πρόταση και έχει προωθηθεί με στόχο να αποφευθεί ο κατακαιρματισμός της ενιαίας αγοράς και για να εξασφαλιστεί η συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα στο υπόλοιπο της οικονομίας μετά την αναθεωρημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή προχωρεί τώρα σε διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας από 11 χώρες μέλη. Όπως είπα, ο κύριος Μοσκοβισή θα είναι στα πιδάλια για το θέμα αυτό. Και σε έφθετο χρόνο βέβαια, θα γίνει ευρύτερη συζήτηση, είμαι βέβαιος, και πέρα από αυτό δεν νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω περισσότερες λεπτομέρειες για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Για τη λεύκανση, για τη λεύκανση του χρήματος. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Με συγχωρείτε. Ναι. Για τον κανονισμό για τη λεύκανση του βρώμικου χρήματος δεν νομίζω ότι μου έγινε πλήρης ενημέρωση τις τελευταίες αυτές δύο εβδομάδες που ασχολήθηκα με το θέμα αλλά η προσέγγιση μου θα ήταν σαφώς ότι όπως προκύπτει, όπως απορραεί από διεθνείς συμφωνίες είναι μεγάλη σημασία να ρυθμι, της ρύθμισης του θέματος αυτού και να γίνει αυτή η ρύθμιση βάσει κοινών κανόνων. Τις λεπτομέρειες όμως δεν είμαι σε θέση να σας εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ και τώρα λοιπόν... Θα... Επ' αυτό θα διεξαχθεί τριμερής διάλογος έτσι κι αλλιώς. Ashley Fox, του ECR. Good afternoon, Lord. Καλησπέρα, Λόρδε Χίλου. Κατά τη τελευταία κοινοβουλευτική θητεία κάποιοι εξημών πέρασαμε πάρα πολύ καιρό και ε, εργαστήκαμε για το Solvency 2. Η καθυστέρηση για την ολοκλήρωση της πρότασης αυτής κόστησε στην ε, χρηματοοικονομικό κλάδο πάρα πολύ και σε χρόνο και σε κόστος. Κόστος που τελικά ε, μετακυλίεται στους καταναλωτές. Οι μοναδικοί που χάρηκαν φαντάζομαι ήταν οι δικηγόροι και οι λιμπίστες. Πότε θα διασφαλίσετε, πώς θα διασφαλίσετε λοιπόν ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για τις συντάξεις δεν θα γίνεται επόμενο Solvency 2 και πώς θα διασφαλίσετε ότι η οδηγία θα λάβει υπόψη την πολύ διαφορετική ε, φύση των συνταξιβετικών συστημάτων και παροχών στα διάφορα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ για απάντηση. Ξέρω ότι η διαδικασία έγκρισης του Solvency 2 ήταν μια μακρά διαδικασία και υπήρξαν και ριζοσπαστικές αλλαγές στι χρηματοπιστικέ αγορές οι οποίες χρειάστηκαν να ληφθούν υπόψη. Το βασικό στοιχείο το οποίο αναφέρεται με βρίσκει σύμφωνο, το συμμερίζομαι. Στα θέματα αυτά όσο πιο γοργά μπορεί κανείς να ανταποκριθεί και να τα επιλύσει και να δώσει σταθερότητα και βεβαιότητα στις επιχειρήσεις και στις εταιρείες προκειμένου να μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους τόσο το καλύτερο. Σε ό,τι αφορά τα, χρηματο... τα συνταξιδοτικά ταμεία και σε ό,τι αφορά τη σχετική οδηγία για τις συντάξεις, αυτό που θα πρέπει να σας καθησυχάζει, αλλά το σημείο κίνησης είναι λίγο διαφορετικό. Η Επιτροπή πριν από το Κοινοβούλιο δεν περιορίζει τις κεφαλαϊκές, κεφαλαϊκές απαιτήσει για την, τις συντάξεις. Η πρόταση αυτή η οποία η αναθεώρηση της οδηγίας του 2003 περιορίζεται στην κυβέρνηση και στην ε, διαφάνεια και τους σχετικούς κανόνες. Πιστεύω ότι αυτό συνάδει με την ε, έκθεση του Κοινοβουλίου του 2013. Για ένα συνδυασμό λοιπόν λόγων πρέπει να σας πω ότι δεν αναμένω αυτή η διαδικασία να διαρκέσει ούτε το μισό από αυτό που πήρε η διαδικασία για το Solvency 2. Θεωρώ ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα για τους φιλελεύθερους, Μάικλ Τόια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, Λόρδι Χίλ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η ρητορία σας και η ευφία σας, αλλά έλλειψη και η έλλειψη ουσία σας. Απαντήστε την ερώτηση που έχουν θέσει δύο συνάδελφοι από τους φιλελεύθερους. Τρία συγκεκριμένα βήματα που θα κάνετε ως Επίτροπος για την εισαγωγή της ε, Ένωσης ε, Κεφαλαίου Αγοράς. Κατά δεύτερον, σας πρότεινε η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους που είναι εκτός της Ευρωζώνης και που ο τραπεζικός κλάδος διοργανώνεται σε εθνικό επίπεδο. Ως Επίτροπος για τα χρηματοδοτικές αγορές θα γνωρίσετε σε βάθος τα τραπεζικά μυστικά των τραπεζών στην Ευρωζώνη. Πιστεύετε ότι από αυτό θα μπορούσε να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων και αν ναι, πώς προτίθεστε να το επιλύσετε. Απάντησε ο Λόρδο Χιλ. Καταρχά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει οποιαδήποτε συμφέρον, σύγκρουση συμφερόντων. Όπω σα είπα και προηγουμένω, θεωρώ ότι βρίσκομαι σε ακριβώ την ίδια θέση όπω ο κύριο Μπαρνιέ. Αλλά αντίστροφη. Για το πώ θα επιλύσω τέτοια ζητήματα, νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι οι δεσμεύσει μου, βάσει των δεσμεύσεών μου, βάσει των συνθήκων και βάσει του όρκου ενώπιον του δικαστηρίου. δεν είναι πράγματα τα οποία κάνει κανείς με ελαφριά καρδιά. Υπάρχει ηθική και νομική υποχρέωση. Αυτή αποτελεί τη βάση επί της οποίας προτίθεμαι να λειτουργήσω και να δράσω σε ό,τι αφορά την Ένωση Κεφαλαίου Αγοράς και σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τα 300 δισεκατομμύρια εδώ και το σχέδιο επένδυσης του Πρόεδρο Γιούγκαρ για τα μακροπρόθεσμα ταμεία επενδύσεων μίλησα. Ένα πλαίσιο πρόληψης για τα προϊόντα της τυλοποίησης για να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας τυλοποίηση και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το δυναμικό ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να καταστούν οι αγορέ αυτές πιο ελκυστικέ. Έχουμε τα εφαρμοστικά μέτρα του MIFID 2, τα οποία θα συμπεριλάβουν τις ε, απαιτήσει και τις προδιαγραφές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό είναι κάτι άλλο. Και επίσης έχουμε να κάνουμε και ένα, με ένα ζήτημα το οποίο άπτεται τον, ε, για τις πιστώσεις σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, μπορεί να υπάρχουν εξέλιξεις, λυπάμαι. Αν δεν έχω ακόμα ένα πλήρες αναπτυγμένο σχέδιο, έχω κάποια στοιχεία, θα επανέλθω όμως. Θα προτιμούσα να τα εξετάσω με την ησυχία μου και να σας προτείνω ένα λογικό σχέδιο για το μέλλον. Ευχαριστώ, Έστερντε για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λόρδο Χίλ, χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα ότι δεν πιστεύετε στην ε, λύση, ότι ε, μία λύση ταιριάζει σε όλους. Ούτε εγώ το πιστεύω, ούτε οι Ολλανδοί, το Ολλανδικό εκλογικό σώμα, θα μας διασφαλίσετε, θα μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι το σύστημα συνταξιοδότησης, το οποίο είναι ιδιαίτερο, δεν θα ε, αναγκαστεί να προσαρμοστεί στα συστήματα άλλων. Κατά δεύτερον, πολλοί συνάδελφοι σας ρώτησαν για την πρόσβαση σε εναλλακτικέ πηγές ε, χρηματοδότησης, ιδιαίτερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χάρηκα που άκουσα τα αρχικά σας σχόλια για τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αναφερθώ στις ε, συνεταιρισμού που αποτελούν συστήματα οργανωμένα από κάτω προς τα πάνω, όπου υπάρχει και δανεισμός στους συνεταιρισμούς αυτούς μεταξύ αγροτών, για παράδειγμα. Και έτσι αποτελείται, αποτελεί αυτό μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. Εσείς μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι θα εξερεχθούν αυτά τα συστήματα εναλλακτικής ε, ε, χρηματοδότησης από ενδεχόμενο από ένα ενδεχόμενο CRD4. Συμφωνώ ιδιαίτερως είναι η απάντηση με την ε, αρχή που κρύβεται κάτω από τα δύο παραδείγματα αυτά που αναφέρατε. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τις μικρές αυτές οργανώσεις, τις συνεταιρισμούς, τις οργανώσεις αυτές, τις οποίες θα πρέπει κατά βάση να ενθαρρύνουμε. Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις για να επανέλθω και στο ερώτημα του κυρίου Φόξ για τη σχετική οδηγία για τις συντάξεις. Νομίζω ότι είναι διαφορετική η προσέγγιση μας συνολικά, αλλά ήδη πρέπει να σας πω ότι ανταλαμβάνομαι το πόσο θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις σε όλους τους τομείς προκειμένου να αναγνωρίσουμε τις διαφορές στις αγορές και να υποβάλουμε λύσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα προς το συμφέρον των εμπλεκομένων φορέων. Thank you. Now, Scott Cato Ευχαριστούμε και τώρα η Μόλι Σκοτ Κάτω από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ. Αναφέρατε στις γραπτές σας απαντήσεις ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της θητείας θα είναι η επαναδιαπομάτευση των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο παρελθόν η Βρετανική κυβέρνηση έχει θέσει ένα αμφιβόλο για πολλά χρηματοπιστωτικά θέματα του ευρωπαϊκού κανονισμού. Περιμένετε μελλοντικέ ε, τέτοιε κινήσει. Ε, και επίση είδαμε πολλέ ερωτήσει για την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων να έχουν τεθεί ω τώρα. Τι θα κάνετε με την επαναδιαγμάτευση του επιδιώκει το Ηνωμένο Βασίλειο και τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με το σύντη του Λονδίνου να είναι μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο τη Ευρωζώνη, εκτό Ευρωζώνη μάλλον, ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώ. Πώς θα λάβετε υπόψη τα παράγωγα, τις ε, κεφαλαίες ε, και όλους τους κανόνες που ισχύουν για τις ασφαλιστικές και ε, εταιρείε και τα τραπεζικά ιδρύματα. Και ως πρώην μέλος της Βρετανικής κυβέρνησης βλέπετε να υπάρχει κάποιος ρόλος στην επαναδιαγμάτευση αυτού του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, κάποιος ρόλος συγκεκριμένο για σας και τι θα γίνει αν υπάρξει ενδεχομένω αντίφαση μεταξύ των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχω μια σχετικά απλή απάντηση σε όλα αυτά. Θέλω να είμαι Ευρωπαίος Επίτροπος. Δουλειά μου θα είναι να αναλάβω τις αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου μου όσο καλύτερα μπορώ βάσει των ικανοτήτων μου. Η οποιαδήποτε επαναδιαπραγμάτευση, η διαδικασία μεταρρύθμισης η συζήτηση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλού και άλλων κρατών μελών είναι κάτι που θα απασχολήσει εκείνους. Αυτή είναι σε κάθε περίπτωση η άποψή μου και δεν βλέπω να υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος. Θα είναι δική μου, θα είναι χαρά μου να φέρω εις πέρα στα καθήκοντά μου ως Ευρωπαίος Επίτροπος. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα για την EFT ο Μάρκο Τζάνι. Ευχαριστώ Κύριε Χιλ, όταν ανακοίνωσε ο Γιούνκερ τον κατάλογο των υποψήφιων επιτρόπων, η επιλογή φάνηκε να είναι ένα έργο πολιτική άπειρα. όπου ο κάθε επίτροπο είχε αναλάβει το πλέον άστοχο χαρτοφυλάκιο και εσεί είστε το πιο αντιφατικό μεταξύ όλων αυτών, όπω είναι ένα Βρετανό παρατηρητή. Το χαρτοφυλάκιο για ε, την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι ένα κόλαφο που δεν μπορεί να δεχτεί αυτό το κοινοβούλιο. Ε, το είπε κάποιο που είναι φίλο των ανάλογων λόμπι. Μάλλον για εσά ότι είστε φίλο των ανάλογων λόμπι. Στη χώρα σα κυριαρχούν ε, συμφέροντα οικονομικά εκτό Ευρωζώνη. Και εσεί είχατε πάντα το πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο των λόμπι και των εταιριών, ενώ θα καλείστε πλέον να διευθετείτε τι κεφαλαίε αγορέ. το ιδιαίτερα δραστήριο στην προάσπιση των συμφερόντων των κερδοσκόπων. Οπότε σα ρωτούμε, μπορείτε να καθησυχάσετε του πολίτε ότι θα, έχετε, θα είστε αμερόληπτο σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα όπω την διευθέτηση των χρηματοπιστωτικών βασικών υπηρεσιών πιστεύει, πιστεύετε ότι αρκεί να πουλήσετε το πακέτο των μετοχών που κατήχατε για να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Είστε ένα πρώην, ε, κάποιο που πρώην είχε συμφέροντα στο χώρο αυτό και τώρα θα προστατεύσετε το χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Σα το λέω γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτε έχουν σοβαρότατε αμφιβολίε. Ευχαριστώ. Κατά πρώτον, όπως είπα, με ρωτάτε για το αν πούλησα το πακέτο των μετοχών μου. Δεν ήταν και τόσο φοβερό αυτό το πακέτο, αλλά οι μετοχές που είχα ήταν μίας εταιρεία δικής μου, οι οποίες πουλήθηκαν. Είπα ότι πούλησα και την εταιρεία μου και πουλήθηκαν σε 24 ώρα μετά τον διορισμό μου στην ε, Βρετανική κυβέρνηση. Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό που μου αποδίδεται ούτε για τον τρόπο με τον οποίο θα φέρω εις πέρα στα καθήκοντά μου, ούτε για την πορεία μου ως τώρα, ούτε για τη χώρα μου παρεπιπτόντος. Όπως έχω πει και προηγουμένως, έχω μια πολύ σταθερή και σαφή άποψη. Και βάσει των συνθηκών και βάσει του επίσημου όρκου μου, αυτή, αυτό το λειτουργήμα δεν το λαμβάνει κανείς ελαφρά την καρδία. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος θα είχα παρατηθεί εάν έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θα φέρω εις πέρα στα καθήκοντά μου προς όφελος του ευρωπαϊκού συμφέροντος Η Κατερίνη Στίλερ τώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιούνκερ θέλει να διασφαλίσει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα λάβει υπόψη και τα συμφέροντα των καταναλωτών και των επενδυτών με τα σχετικά μέτρα που θα βελτιώσουν τη θέση των πολιτών. Σύμφωνα με τις στατιστικές, μόνο 25% των πολιτών εμπιστεύονται τις τράπεζες. Θα συμφωνήσετε ότι είναι μικρό το ποσοστό αυτό. Ποια βήματα προτίθεστε να λάβετε για να επαναφέρετε την εμπιστοσύνη των πολιτών στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, να τα κάνετε αυτά πιο διαφανή και πιο ανταγωνιστικά και να διασφαλίσετε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών οριζόντια. Και σύμφωνα και με την πλέον πρόσφατη ε, νομοθεσία. Απάντηση. Δεν έχει μικρόφωνο νομίζω. Μάλιστα. Νομίζω ότι θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα και όπως νομίζω είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, το να στοχεύσει κανείς την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών για τα επόμενα πέντε χρόνια είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς τα τελευταία πέντε χρόνια η ικανότητα του συστήματος των υπηρεσιών της παρούσας επιτροπής χρειάστηκε να δοθούν όλες οι προσπάθειες δηλαδή για την διάσωση του συστήματος. Έχοντας την κρίση πίσω μας τώρα μπορούμε να διαθέσουμε περισσότερο χρόνο και περισσότερες προσπάθειες στο να σκεφτούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα πλεονεκτήματα σε καταναλωτές και πολίτες. Και αν το δει κανεί από την πρακτική σκοπιά, για παράδειγμα ασφαλιστικά προϊόντα, αυτοκινήτων, σπιτιών, που ποικίλουν πολύ από αγορά σε αγορά και ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν πολύ περισσότερα σε κάποια τμήματα της αγοράς από ό,τι άλλο. Η ε, καθυστερή για παράδειγμα η καταβολή της ε, ασφαλιστικής αποζημίωσης. Νομίζω ότι αν βρούμε πραγματικούς, πρακτικούς τρόπους να προσφέρουμε όφελος, πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν, με περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη πληροφορία, τα... την ενημέρωση του καταναλωτού να γνωρίζει για ποιο πράγμα υπογράφει. Πρέπει να αναζητήσουμε και άλλους τρόπους να αναπτύξουμε τα πράγματα αυτά. και οι προμήθειες που λαμβάνουν οι φορείς προσφοράς υπηρεσιών. Να γνωρίζεις δηλαδή τι πληρώνεις και τι λαμβάνεις. Καλύτερο παρά να είναι ασαφές και να μην γνωρίζεις γιατί κάποιος σου πωλεί το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι πλούσιος ο τομέας αυτός, πολύ ευχαρίστως θα δεχθώ ε, προτάσεις και από την Επιτροπή σας Προστασία Καταναλωτών αλλά και από άλλους για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ευχαριστώ πάλι και η η ECR. Ευχαριστώ, Lord Hill. Μου δίνετε την ευκαιρία να θέσω δεύτερη ερώτηση. Θα έρθω στα τεχνικά θέματα που μας έχουν απασχολήσει τα τελευταία πέντε χρόνια στην Οικονομική Επιτροπή και ιδιαίτερα μέσα στα, πλαίσια των νομοθετημάτων που ε, έχουμε ε, συζητήσει είχαμε και το τα καθεστώτα τρίτων χωρών που αμφισβητήθηκαν συχνά. Αυτά τα θεωρείτε, θεωρείτε ότι πρέπει να υπαχθούν σε μια συνολική όμνιμπους οδηγία. όπως Εμίρ, Μιφίντ και άλλες αγορές που έχουν ειδικά καθεστώτα. Πάντα ε, μέσα σε αυτά τα διεθνή πλαίσια είπατε για την ε, επίλυση για την εξυγεία των τραπεζιών και για τα CCDs. Αυτό εκεί να μου πείτε κάτι. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε. Σχετικά με μια συνολική οδηγία. Δεν το ε, συζήτησα βέβαια μέσα στην ενημέρωσή μου των δύο τελευταίων εβδομάδων, αλλά είναι κάτι το οποίο αξίζει να μελετηθεί. Η γενική μου προσέγγιση, όπως είπα και πριν, σε ό,τι αφορά την προσέγγιση στην νομοθεσία, θα είναι να προσπαθήσω να εξασφαλίσω μια συνοχή των δράσεών μας σε έναν αριθμό τομέων. Βεβαίως και λόγω του τεχνικού χαρακτήρα, αλλά και λόγω του όγκου των δράσεων και του γεγονότος ότι πολλά προέρχονται από διαφορετικές νομοθετικές βάσεις και να δούμε πώς διασυνδέονται οι διάφοροι τομείς της νομοθεσίας μεταξύ τους. Αυτό είναι δύσκολο. Και γενικό κανόνα, νομίζω που ισχύει, είναι ότι όσο πιο απλέ είναι κάποιε ρυθμίσει, τόσο καλύτερα. Βεβαίω αυτά που λέτε θα τα διερευνήσω και θα δω εάν υπάρχει κάποια αξία στην ιδέα αυτή ή όχι. Γενικότερα τώρα, για το Central Counterparty Clearing. Η κατάσταση όσο έχει σήμερα δεν είναι ικανοποιητική. Χρειάζεται να βρεθεί μια διαρκής λύση. Γνωρίζομαι ότι πρόκειται για μια πρόκληση που πρέπει να λύσουμε. Καλά θα είναι να μπορέσουμε να παράσχουμε ισοτιμία στους Αμερικανούς, αλλά θα πρέπει και αυτοί να μπορούν να αναφέρονται περισσότερο στους δικούς μας κανόνες. Γνωρίζω ότι επ' εργαζόταν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρνιέ και εγώ θα ακολουθήσω την πορεία που έχει χαράξει. Ματ Επανέρχομαι κύριε Επίτροπε στην σύγκρουση συμφερόντων. Θα γνωρίζετε ότι πολλοί σχολιαστέ και ευρωβουλευτές παρόντες εδώ εξέφρασαν την ανησυχία ότι διαθέτεται επενδυμένα συμφέροντα στο ΣΥΡΙ του Λονδίνου όπου έχετε αναπτύξει τα επαγγελματικά και προσωπικά σας δίκτυα. Παρακολούθησα και ορισμένους υποστηρικτές σας εδώ που εξέφραζαν την ελπίδα ότι θα στηρίξετε την μείωση των νομοθετικών ρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Εγώ δεν συμφωνώ ότι λιγότερη ρύθμιση είναι και καλύτερη. Θέλω λοιπόν να σας ερωτήσω, ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις θεωρείτε ότι πρέπει να επανεξεταστούν. Θεωρείτε ότι ορισμένε πρέπει να ενισχυθούν. Και τελευταία ερώτηση. Πώς προτίθεστε να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη των πελατών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Πώς θα δώσετε προτεραιότητα στην προστασία των δικών τους συμφερόντων απέναντι σε ένα κλάδο που πολλοί ισχυρίζονται ότι έχετε πάρα πολλές στενέ διασυνδέσει μαζί του. Ας ξαναπώ τα ίδια. Πριν από μια-δυο ερωτήσει, είπαμε πόσο σημασία έχει να σκεφτούμε καλά τα συμφέροντα των πελατών και καταναλωτών και αυτοί να ωφεληθούν τελικά. Αυτό θα ήθελα να κάνω. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά τη γενική προσέγγιση, στην νομοθεσία. Είπατε, νομίζω ότι δεν συμφωνείτε ότι λιγότερη ρύθμιση είναι και καλά καλύτερη. Α, θα σας τρομάξω, αλλά συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται το σωστό ποσό ρύθμισης. Είδαμε όμως και τι έγινε όταν δεν υπήρχε επαρκής ρύθμιση. Μην μου αποδώσετε λοιπόν απόψεις που δεν έχω σχετικά με την σημασία της νομοθεσίας και σχετικά με την αποκατάσταση σωστής ισορροπίας ανάμεσα σε μια νομοθεσία που να λειτουργεί και σε μια αγορά που να λειτουργεί. Δεν είπα και δεν λέω και ούτε πιστεύω ότι χρειαζόμαστε να ρίξουμε στην πυρά τα πάντα. Αυτά που χρειαζόμαστε είναι να εξετάσουμε λογικά και ρεαλιστικά τις ρυθμίσεις που έχουμε θεσπίσει και έχουμε ούτως ή άλλως ένα σύστημα αναθεώρησης της, νομολογίας, της ε, νομοθεσίας μέσα στα ε, πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας. Αλλά εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε και τη σωστή ισορροπία. Και ο λόγος είναι ότι αν εξετάσετε οποιονδήποτε τομέα, που μπορώ να σκεφτώ εγώ τουλάχιστον, όπου κάποιοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια κρίση με μεγάλη ταχύτητα και κάτω από μεγάλη πίεση, όλοι κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά δεν σημαίνει ότι πετυχαίνουν πάντα απόλυτα το στόχο. Σε ό,τι αφορά το City του Λονδίνου, η εικόνα που σκιαγραφείτε δεν την αναγνωρίζω. Άφησα την επιχείρησή μου εδώ και μια πενταετία. Δεν βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος του City του Λονδίνου. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Φιλίπ Ντεμπάκερ των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κάποια πράγματα ακόμη δεν έχουν αποσαφενιστεί προφανώς. Η πρώτη με ερώτηση, και θα ήθελα μια απλή μονολεκτική απάντηση ναι ή όχι, είναι για την Τραπεζική Ένωση. Θα προβλέψετε τον τελικό πυλώνα, δηλαδή το πρόγραμμα εγγύηση των καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα στο 12 μήνο μετά την ανάληψη καθηκόντων, ναι ή όχι. Και έπειτα πέραν από το σύστημα που έχουμε για τι μεσαίε και μικρομεσαίε επιχειρήσει και την ε, προστασία του, δεν δώσατε πιστική απάντηση, διότι εδώ ο ερευνητικό ρόλο τη νομοθεσία παίζει σημαντικό ρόλο. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι συγκεκριμένη. Ποιε ήταν οι προτεραιότητέ σα, θα άρετε κάποιε από, ε, ε, από του φραγμού όπως το MIFID, το Solvency 2, το MIFID 2 για τις, ε, για τις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τα IBO. Η, η αγορά IBO ε, δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη επαρκώς. Τι θα κάνετε λοιπόν για τις εταιρείες ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά μετοχών και να μπορούν να βελτιώσουν την κατάστασή τους. Θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις για αυτές τις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτον, για την Τραπεζική Ένωση δεν είμαι σε θέση να σας δώσω απάντηση διαφορετική από αυτή που έδωσα τουλάχιστον μία ή δύο φορές προηγουμένως για το πρόγραμμα εγγύησης των μεταθέσεων. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να απαντήσω με ναι ή όχι. Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργήσει και μετά είναι το χρόνο, ως συνήθως, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικό και αν χρειάζονται αλλαγέ. Θα ήθελα να μπορώ να απαντήσω, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα θέλατε. Ως προς την Ένωση Κεφαλαίου Νομίζω τα παραδείγματα που δώσατε και τους φραγμούς που θα θέλαμε να υπερβούμε, νομίζω εδώ αυτός είναι ένας από τους πολλούς τομείς όπου θα πρέπει να δράσουμε. Αλλά μετά από δύο μόλις εβδομάδες και προτού εφόσον να γίνεται, αναλάβω τα καθήκοντά μου, δεν είμαι στο επίπεδο γνώσης λεπτομεριών για να σας πω αυτός ο κανονισμός πρέπει να αλλάξει έτσι και να καταργηθεί ο άλλος και να προτείνω τον εξή νέο. Θα πρέπει να δούμε όλους αυτούς τους φραγμούς εφόσον τους εντοπίσουμε και μετά να εξεύρουμε μια πρακτική απάντηση για πράγματα που θα πρέπει να αλλάξουν, για πράγματα που θα πρέπει ενδεχομένω να εισαχθούν. Το rule book, οι κανόνες θα πρέπει να διευρυνθούν, να, να διορθωθούν. Αυτό θα ήθελα να το δω μαζί σας και με όλους όσοι έχουν ιδέες για το θέμα αυτό. Είναι ανοιχτή η συζήτηση, δεν έχει ολοκληρωθεί και πέραν αυτού Σύντομα θα προκύψει και το χρονοδιάγραμμα με πολύ συγκεκριμένο πλάνο δράσης. Θα ξεκινήσουμε γρήγορα με κινήσεις για να δώσουμε κίνητρα για την υψηλή επιπέδου και υψηλής ποιότητας τιτλοποίηση και μετά βήμα το βήμα θα